Ορίστε, καλημέρα. Ξέρω ότι είναι νωρίς για σας, αλλά... Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε, γιατί αλλιώς... Αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο. Είναι 9 και 4. Αλλά δεν έχουν όλη την ίδια ώρα βέβαια, τι να κάνουμε. Ας πούμε ότι είναι 9. Γιατί τα ορολόγια εδώ είναι γνωστό ότι καθυστερούν. Λοιπόν, έχουμε μια ώρα για κάθε για τον Στίβεν Μάγερ καταρχήν και οι ερωτήσεις θα ακολουθούν τις συνήθεις αρχές. Ένα λεπτό για την ερώτηση και 3,5 λεπτά για την απάντηση. Σύνολο 5. Παρακαλώ τους βουλευτάς να θέτουν ένα ερώτημα, όχι πολλαπλά. Αλλιώς θα απαντά ο υποψήφιος μόνο στη λογικότερη από τις πολλαπλές ερωτήσεις. Καταρχήν λοιπόν ο Στέφανος Μάγιορ θα έχει πέντε λεπτά για να κάνει ορισμένες προκαταρκτικές δηλώσεις και μετά θα γίνουν οι ερωταπαντήσεις. Σας ε, υπενθυμίζω ότι είναι ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Αγορών κλπ. Ορίστε Στέφανε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την εισηγήση σε αυτήν και ευχαριστώ και τα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής που μου δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε. EU structure η θέση την οποία φιλοδοξώ να καταλάβω είναι από τις σημαντικότερες για την αντιμετώπιση της κρίσης. Έχουμε καταλάβει και δύσκολα κιόλα ότι χρειάζεται κάποια δημοσιονομική επιτήρηση η οποία σε καθαρά εθνικό επίπεδο δεν λειτουργεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο στον καθορισμό αυτού του νέου επιτηρητικού πλαισίου, εποπτικού πλαισίου και τώρα αναμένει πολλά. Επομένως, για την αντιμετώπιση επιγόντων καταστά... επιγουσών καταστάσεων κυρίως χρειάζεται η θέση αυτή που τη λέμε έσμα μεταξύ μας. Θα ήθελα λοιπόν να, να τονίσω πέντε προτεραιότητες μου. Πρώτη, μία πραγματική εποπτεία κινητών αξιών κλπ. Ο ρόλος εδώ της ΕΣΜΑΣ θα είναι οι υπάρχουσες πρακτικές επιτήρησης να συμφωνούν με τις ε, αρχές που θα έχουν τεθεί και με ό,τι προκύψει ως ανάγκες. Δεύτερη προτεραιότης, η προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών. Σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές και οι καταναλώτες και μάλιστα οι δημοσιονομικοί καταναλωτές δεν την χάνουν των υπηρεσιών που τους αξίζουν. Εδώ ο ρόλος της ΕΣΜΑΣ λοιπόν θα είναι απλότης και διαφάνεια. Ας πούμε προειδοποίηση βλαβερών προϊόντων ή και απαγόρευσή τους. Τρίτη προτεραιότης. Συμβολή στη σταθερότητα. Η ΕΣΜΑ δεν θα είναι απομονωμένο όργανο αλλά τμήμα ολόκληρου πλαισίου. Θα συνεργάζεται δηλαδή με κάθε τραπεζική και ασφαλιστική αρχή και με άλλες ευρωπαϊκές αρχές για να κάνει συστάσεις και να τις εφαρμόσει όταν χρειάζεται. Τέταρτη προτεραιότης, ενιαίοι κανόνες και πρότυπα. Και πέμπτη, το ισόπεδο γήπεδο όπως λέμε πολλοί από εμά για την επιτήρηση, για την υποπτία. Η ΕΣΜΑ πρέπει να έχει τη δικαιοδοσία να δράσει όταν παρατηρεί ότι μπορεί να έχει παραβιαστεί το κοινοτικό δίκαιο. Αυτές οι πέντε προτεραιότητες είναι η βάση του προγράμματος δράσης της ΕΣΜΑ για την επόμενη περίοδο είναι φανερό ότι η αλλαγή από τον Κέσαρα στο ΕΝΕΣΜΑ θα είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό ποιοτική αλλαγή και διοικοδοσίες αλλαγμένες και με το μέγεθος της υπηρεσίας και η ποιότητα των εργασιών της. Τέλος. Τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να τεθώ επικεφαλής δύο ανάλογων οργανισμών. Ο πρώτος ήταν η Ολλανδική Αρχή Κινητών Αξιών και η δεύτερη η ΕΣΚΟ. Από τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρα στις δύο αυτές θέσεις είναι ότι η ανεξαρτησία είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός επόπτη η οποία απαιτείται και για τη θέση αυτή η δράση μου θα συμβάλλει στη σταθερότητα από την άλλη της ευρωπαϊκής αγοράς κινητών αξιών. Τέλος, είμαι υπόλογος προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το οποίο όπως είπα και νωρίτερα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να φτάσουμε μέχρι εδώ για τον καθορισμό αυτής της αρχής δηλαδή. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι και στο μέλλον θα παίξει σημαντικό ρόλο η δράση της ΕΣΜΑ, της ΕΑΚΑ δηλαδή. Και ως πρόεδρος της θα επιζητήσω διάλογο με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ καλή αρχή. Περίσσεψαν και 15 δευτερόλεπτα. Ο πρώτ, η πρώτη ερώτηση είναι από τον Ζαν Πολ Γκοζές, εκ μέρου του ΕΛΚ. Ζαν Πολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιο Πρόεδρε, τα λόγια σας ήταν πάρα πολύ συμπαθή και ευχάριστα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που όπως είπατε έκανε πολλά για να επιτύχει την ευρωπαϊκή εποπτεία. Όλα όσα είπατε ε, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλά. Δεν αμφισβητώ το πρόσωπό σας, αλλά θα σας πω ειλικρινά ότι κάποιοι από εμά αμφισβητούμε την ε, δυνατότητα που θα έχει η ΕΣΜΑ να θέσει σε εφαρμογή τις αρμοδιότητες τις οποίες τις αναθέτουν ε, ο κανονισμός. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι επιλογές, η επιλογή της ιεραρχίας οδηγούν στο να έχουμε έντονους φόβους πως δεν θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ΣΥΖΑΡ και την ΕΣΜΑ. Έχουμε πολύ μεγάλες λοιπόν αμφιβολίες ως προς αυτό. Μπορείτε ενδεχομένως να μας δώσουμε κάποιους βάσιμες λόγους που να άρουν αυτές τις αμφιβολίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω την διαφορά ανάμεσα στην προηγούμενη κατάσταση με την Caesar και τη νέα κατάσταση με την ΕΣΜΑ. Θα ήθελα να τονίσω ότι μια σημαντική αλλαγή είναι η αρμοδιότητα που ανατίθεται στην ΕΣΜΑ μέσω του κανονισμού. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι, οι, οι οργανισμοί αξιολόγησης θα είναι υπό την άμεση υποπτία της ΕΣΜΑ. Θα, αυτό είναι διαφορετικός ρόλος τελείως από την ΣΥΖΕ. Δεν είχε τέτοιο ρόλο η ΣΥΖΑ, δεν μπορούσε άμεσα να υποπτεύσει οποιοδήποτε οργανισμό. Ένα παράδειγμα θεμελιώδους αλλαγής λοιπόν. και σε άλλους τομείς υπάρχουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Δηλαδή η δυνατότητα να θέσει προδιαγραφές ε, σε συνεργασία με την Κομισιόν και εκεί παίζει ρόλο και το Κοινοβούλιο και η δυνατότητα να ενεργήσει σε περίπτωση ρυθμιστικού ανταγωνισμού. Όσον αφορά λοιπόν τις αρμοδιότητες της ΕΣΜΑ υπάρχει σαφής διαφορά από το παρελθόν και δεν θα είναι σταδιακή αλλαγή εκεί αλλά θεμελιώδης αλλαγή, ρηξικέλευθη. Επίσης όσον αφορά το σπόρους ε, που διατίθενται στον οργανισμό θα είναι διαφορετικό το μέγεθος. Ήταν 40-50 άνθρωποι μόνο παλαιότερα, ενώ στα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν πάνω από, θα γίνουν πάνω από 100. Νομίζω ότι και αυτό θα παίξει, θα παίξει ρόλο και θα έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ε, αρμοδιότητες, πόροι, ηγεσία. Θα είναι πολύ διαφορετικός οργανισμός. Αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι εύκολο να δημιουργηθεί αυτός ο νέος οργανισμός. Αλλά όσον αφορά τους πόρους, αν συναντήσω προβλήματα ως πρόεδρος, θα σας τα αναφέρω και θα είναι ξεκάθαρα όλα αυτά τα θέματα. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος είναι ο Ούντο Πούλμαν, εκ μέρους των, ε, της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε εδώ στην Επιτροπή, κύριε Μάιτζορ. Θα κατανοείτε ασφαλώς ότι η Επιτροπή αυτή και αυτό το Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερο υπερήφανα που έχουμε μια ιδιαίτερο ε, δευμεσμένη νομοθεσία όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και την πετύχαμε. Βεβαίω θέλουμε στην κορυφή αυτών των νέων εποπτικών οργάνων να δούμε κάποιου ανθρώπου που πραγματικά ε, ε, προσπαθούν για την ενίσχυση αυτού του πνεύματο, ούτω ώστε να υπάρχει μια τέτοιου είδου δέσμευση στην κατεύθυνση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το ερώτημά μου, ε, πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια είχαμε ήδη τις αρμοδιότητες της ΕΣΜΑ. Εάν ήσασταν σε αυτή τη θέση πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, πώς θα τις αξιοποιούσατε, τι θα κάνατε στις συγκεκριμένα, στις συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει υπερβολική ρύθμιση, άλλοι παραπέμπουν στην ε, ε, νομολογία Μερώνη. Εσείς τι θα κάνετε διαφορετικά και τι αναμένετε για το μέλλον. Είναι δύσκολο βεβαίως να πάει κανείς ε, πίσω και να προσπαθήσει να φανταστεί τι θα συνέβαινε εάν η ΕΣΜΑ είχε συσταθεί πριν από την κρίση. Και υποθέτω ότι η υπόθεση είναι ότι τι θα συνέβαινε εάν ε, είχε δημιουργηθεί η ΕΣΜΑ σε μια πρεμότερη φάση. Καταρχήν θα έλεγα ότι η ρυθμιστική εποπτεία δεν συνιστά μια εγγύηση. Βεβαίως θα υπάρχουν ε, κάμψεις στην οικονομία και ακόμα και αν υπάρχει υποπτία δεν, θα, δεν είναι μια εγγύηση για την άφηση της αγοράς. Ωστόσο θα έλεγα ότι η, ότι κανείς δεν ανέμενε ότι θα καταλήγαμε σε αυτή την κατάσταση. Τι θα συνέβαινε λοιπόν εάν η ΕΣΜΑ είχε δημιουργηθεί σε μια προηγούμενη φάση. Νομίζω ότι θα είχε μειώσει ουσιαστικά τους κινδύνους να επισέλθηκαν σε μια τέτοια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Και νομίζω ότι θα ήταν σόφρον να είχαμε εκείνη την εποχή τις εξουσίες που τώρα δίδονται στην ΕΣΜΑ. Όπως είπα προηγουμένως, οι οίκοι αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την κρίση. Υπήρχαν πολύ σημαντικά ποιοτικά θέματα όσον αφορά την αξιολόγησή τους και αν είχαμε πιο νωρί μια τέτοιου είδου εποπτεία, νομίζω ότι αυτό θα κατέληγε σε καλύτερη βαθμολόγηση. Τώρα, όσον αφορά τη ρυθμιστική αρμοδιότητα, ως ε, ρυθμιστής της κάτω χώρας, εγώ είχα το μερίδιό μου σε αυτό τον ανταγωνισμό όσον αφορά τη ρυθμιστική αρμοδιότητα, όπου ε, λέμε σε κάποιον προμηθευτή ότι δεν επιτρέπεται να παράσχει κάποιες υπηρεσίε εφόσον δεν εκπληρώνει τις ε, προδιαγραφές διαφάνειας. Ε, ωστόσο, παρόλα αυτά, μερικές εβδομάδες μετά το ίδιο προϊόν εγκρίνεται σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και προσφέρεται εντό Ευρώπη. Συνεπώ, λοιπόν, ο ρυθμιστικό ανταγωνισμό είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί κατά το παρελθόν και πιστεύω ότι η ΕΣΜΑ έχει δυνατότητα να δουλέψει πάνω σε αυτό. Η... Ε, Επίση, ε, σε εκείνη τη φάση δεν είχαμε διαφάνεια όσον αφορά την αγορά των εξωχρηματιστηριακών παραγόγων. Είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένα από τα αίτια που συνέβαλαν σε αυτή την κρίση. Άρα λοιπόν και πάλι θα έλεγα ότι η ρύθμιση δεν είναι μια εγγύηση 100% αλλά πιστεύω ότι το να έχει κανείς εποπτεία μόνο σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχει την ευρωπαϊκή συνιστόσα γιατί γνωρίζουμε ότι οι αγορές αυτές είναι ευρωπαϊκές είναι ε, δεν θα ε, λειτουργήσει. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θα ήθελα να συνοψίσω σε αυτό το σημείο λέγοντα ότι αν είχαμε την αίσθημα σε μια προηγούμενη φάση, νομίζω ότι θα είχαμε λιγότερε πιθανότητε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε τώρα. Βεβαίως, τμήμα αυτή τη κρίση προέρχεται από, έξω από την Ευρώπη, από άλλε περιοχέ του κόσμου, αλλά και πάλι πιστεύω ότι οι πιθανότητε ότι θα καταλήγουμε σε μια τέτοια είδου κατάσταση θα ήταν πολύ πιο περιορισμένε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούμε την, την ε, μορφή του μιας, ε, του ενός λεπτού για την ερώτηση και με τριάμιση λεπτά για την απάντηση. Γκούλαντ, εξ ονόματος της... Ε, άλτε, Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε συνάδελφοι. Σας είπαν πόσο σκληρά δουλέψαμε εδώ για τη δημιουργία αυτών των αρχών ε, στις γραμμές της έκθεσης Λαροζιέρ. Εγώ έχω να σας θέσω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και μάλιστα προέρχεστε από μια χώρα που πάντοτε ήταν πολύ προσιλωμένη στην εσωτερική αγορά. Το μόνο που κάναμε εδώ είναι να αυξήσουμε το επίπεδο μάλλον να, φέρουμε το επίπεδο των αρχών και των ρυθμίσεων στο επίπεδο που ήδη είχαν φτάσει οι αγορές λόγω της διασύνδεσης τους. Αν ωστόσο υπάρξει κατάχρηση, πράγμα που μπορεί να υπάρξει, η ρήτρα την ρήτρα διασφάλισης που έχει βάλει το Συμβούλιο στο κείμενο, τι θα κάνετε. Well, I would like to express that, uh, Εγώ θα ήθελα να σας πω η ότι η, η ρήτρα η ασφαλιστική δικλίδα μάλλον, η ασφαλιστική ρήτρα αφορά βασικά τα θέματα φορολογίας. Όμως έχουμε και τον τομέα των τραπεζών. Εκεί είδαμε πως τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιήθηκαν για να σωθούν, να διασωθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ήταν, ε, αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα κέριο για τον τομέα των τραπεζών. Για τον τομέα του ΕΣΜΑ να σας πω ότι εγώ έως εξής κατανοώ αυτή τη ρήτρα. Ότι δηλαδή ο ρυθμιστής της ΕΣΜΑ δεν μπορεί να λάβει απόφαση για την ε, χορήγηση, και την κατανομή μάλλον των χρημάτων των ε, φορολογουμένων για την ε, διάσωση. μακροπρόθεσμα οι ρυθμιστές στην ουσία υπάρχουν για να εξασφαλίζουν την ευημερία των αγορών όχι για να τις κάνουν λιγότερο επιτυχής οι ρυθμιστέ αυτό φροντίζουν, ώστε να είναι επιτυχεί οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η ρυθμιστική εποπτεία ώστε να εξασφαλίσουμε πως ε, θα είναι επιτυχής οι αγορές ε, και θα δημιουργηθεί αυτή η βάση, η πιο μακροπρόθεσμη. Ε, η δική μου λοιπόν ερμηνεία αυτή τη ρήτρας ασφαλείας είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση όπου για παράδειγμα δεν δίνεται άδεια και μπορεί κανείς να πει ότι αυτό έχει κάποιο, κάποιο αποτέλεσμα στις αγορές. Εγώ το βρίσκω αυτό ως ένα αντίβαρο στην ε, άλλη λύση όπου θα χρησιμοποιούσε κανείς άμεσα τα χρήματα του φορολογουμένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ο Σφέν Γκίγκαλτ. Γεια σας. Συγγνώμη που άργησα, αλλά έπεσα σε μποτιλιάρισμα. Το Κοινοβούλιο μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο έδωσε <coughs> και στις τρεις αυτές τις ευρωπαϊκές αρχές το δικαίωμα να περιορίζουν κάποιες συναλλαγές, κάποια είδη μάλλον συναλλαγών. Υπό ποιες ε, προϋποθέσεις μέσα στο πλαίσιο της εντολής σας ε, ε, και υπό τις αρμοδιότητες της ΕΣΜΑ θα χρησιμοποιούσατε αυτή τη δυνατότητα. Βλέπετε κάποιο είδους πρακτικές, κάποια είδη προϊόντων που θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν να τα βγάλετε από την αγορά. Ποια θα ήταν τα κριτήριά σας λοιπόν, ποιο θα ήταν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όπου τουλάχιστον θα ξεκινούσατε μια τέτοια έρευνα για το κατά πόσο ε, αυτές οι πρακτικές ε, είναι τέτοιου τύπου. Κοιτάξτε, όπως τόνισα στην ε, εναρκτήριά μου δήλωση, ένας από τους τομείς εστιασμού θα είναι η προστασία του καταναλωτή και η, και η λιανική πώληση. ρόλος μας είναι η προειδοποίηση για την επικινδυνότητα του προϊόντος. Είναι κάτι που έχω κάνει συχνά στι κάτω χώρε, που είχαμε για παράδειγμα ένα, προ, πρόγραμμα το οποίο κερδοσκοπούσε για τις γέ, yes. yes. Δηλαδή αυξάνονταν και μειώνονταν οι τιμές των γεών ανάλογα με τις αγορές που γίνονταν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα ως καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγούμε τους κινδύνους για κάποια προϊόντα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις φαντάζομαι πως όντως θα χρειαστεί να απαγορευθούν κάποια προϊόντα. Ε, αυτό είναι όμως νέο, κάτι καινούριο σε κάποιο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, στη ζωή μου ω ρυθμιστή, το έχω κάνει και παλιότερο που, για παράδειγμα, δεν δίναμε άδεια για κάποιον προμηθευτή όταν είχε κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σχέδιο επιχειρηματικό που μπορούσε κανεί να δει ότι αν ο καταναλωτή αγόραζε το προϊόν στο 70, 80, 90% της προκαταβολής του καταναλωτή. Αυτό δεν θα ήταν η επένδυση, αλλά θα ήταν διοικητικό κόστος ε, ε, και διάφορα άλλα, και διάφορες άλλες τέτοιε δαπάνε. Ποιοι θα ήταν λογικοί λοιπόν υποψήφοι, θα ήταν τέτοιου είδου προϊόντα όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο καταναλωτής να μην είναι ικανοποιημένο με το προϊόν, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει και στις προτιμήσεις του καταναλωτή. Είναι εξαιρετική περίπτωση διότι οι κατανοητέ θέλουν να έχουν επιλογή και να ναι. βλέπουν καινοτομία, άρα πρέπει κανείς να προσέχει όταν εφαρμόζει αυτό το μέτρο. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα όπου και οι προμηθευτέ δεν τα επιθυμούν αυτά τα προϊόντα. Στη χώρα μου υπήρξαν περιπτώσεις και ξέρω και ότι σε άλλε χώρε υπήρξε παρόμοιο παράδειγμα όπου η χρηματοπιστωτική βιομηχανία ολόκληρη είχε πρόβλημα για την παροχή κάποιων ε, προϊόντων και οι καταναλωτές ε, έλαβαν ε, αντιστάθμιση, αποζημίωση για προϊόντα τα οποία μάλιστα αποσύρθηκαν από την αγορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ECR, η Κέι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πάλι θα ήθελα να σας συγγνώμη που ήρθα αργά. Ε, συζητούσαμε την Κομισιόν το όλο πρόγραμμα MIFID και την αναθεώρησή του. Ε, βεβαίως έχουμε, είναι προφανές ότι έχουμε ε, τα προβλήματα των αγορών σε σχέση με τη νέα νομοθεσία που επίκειται και προσπαθούμε να κάνουμε μια αναθεώρηση της MIFID ε, σε σχέση με την αγορά ιδιωτικών επενδύσεων. Νομίζω ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και άλλοι μιλητέ αναφέρθηκαν στο τι έχετε μπροστά σας. Η Σίζαρ εργάστηκε συνεργάστηκε με εθνικές ομάδες. Μπορείτε να μας πείτε ε, κάτι για τις επίσημες ε, συμφωνίες σε σχέση με την στελέχωση των, της ομάδας ρυθμιστών σε εθνικό επίπεδο ε, και τι θα γίνει με τις ε, βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ε, αέρα. Πώς θα συντονίσετε τη δική σας δραστηριότητα με την ΕΣΜΑ. Πώς θα συντονίσετε τις δραστηριότητες της ΕΣΜΑ με τους άλλους ρυθμιστές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές είναι δύο ερωτήσεις Καταρχήν, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη ερώτηση εν σχέση με τις συμφωνίες με τους εθνικούς ρυθμιστές και τη δική τους πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με συγκεκριμένες αγορές. Μεγάλο τμήμα της εργασίας της ΕΣΜΑ θα είναι άμεση εποπτεία. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής εποπτείας θα γίνεται σε εθνικό επίπεδο, όπως το είπα προηγουμένως και η ΕΣΜΑ θα, θα δημιουργήσει τις, τους δικούς τους οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, θα υπάρχει πραγματογνωμοσύνη σε άλλους τομείς, όπου η ΕΣΜΑ θα δραματίζει έναν άμεσο ρόλο εποπτείας. Τώρα, όσον αφορά για αυτού του τομεί, όπου δεν θα ασκείται καθημερινή υποπτή εκ μέρους της ΕΣΜΑ, ε, βεβαίω η εμπειρογνωμοσύνη θα είναι σημαντικό να προέρχεται από του εθνικού ρυθμιστές, από τι χώρε μέλη. Και νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα εδώ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αντιλήσουμε αυτέ τι πληροφορίε και την εμπειρογνωμοσύνη για την ΕΣΜΑ. Ε, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτούς τους οργανισμούς έχουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με την ε, ΕΣΜΑ και να υπάρχει λοιπόν αυτή η ροή εμπειρογνωμοσύνης από το εθνικό επίπεδο στο επίπεδο της ΕΣΜΑ. Και εγώ είμαι ως ο ψήφιος πρόεδρος, είμαι σίγουρος ότι οι εθνικοί ρυθμιστές θα ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με τη δική τους εμπειρογνωμοσύνη στην ΕΣΜΑ. Έπειτα θα υπάρχουν διάφορες επιτροπές οι οποίες θα παίζουν ένα ρόλο σαν αφορά την παροχή συμβουλών, ε, τις συστάσεις, διατύπωση συστάσεων και την ανάπτυξη των ε, τεχνικών προδιαγραφών θα υπάρχει ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστών και τέλος ε, σε κάποιο... Ε, και ε, βαθμό βέβαια θα ασκεί και το ρόλο της ΕΣΜΑ. Ωστόσο θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΣΜΑ θα είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός και θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική της βάση εμπειρογνωμοσύνης. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία όσον αφορά την άντληση εμπειρογνωμοσύνης από, τα, από τις χώρες μέλη, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μια βασική ομάδα η οποία να δημιουργεί την εμπειρογνωμοσύνη στις χρηματοπιστωτικές, σχέση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τώρα, όλες οι εξουσίες όσον αφορά το συνολικό πλαίσιο και το ρόλο της ΕΣΜΑ στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι ένα από τα σημεία τα οποία έθεσα στην ενακτήριο ομιλία μου αφορά τον ρυθμιστικό ανταγωνισμό. Και θα ήθελα να καταστήσω ρητό ότι ένα από τα αίτια αυτής της κρίσης ήταν ο ρυθμιστικός ανταγωνισμός. Στην ε, Ευρώπη συνέβη κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι βεβαίω ο αριθμιστικό ανταγωνισμό να μην συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, η συνεργασία στο επίπεδο των G20 είναι ιδιαίτερο σημαντική και πολλά μέτρα συντονίζονται σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό το διαπιστώνουμε. Επίση υπάρχει ένα ειδικό ρόλο για την ΕΣΜΑ. Δώσατε το παράδειγμα τη SCC η οποία δεν διατυπώνει μόνο τις προδιαγραφές αλλά εποπτεύει και τις αγορές και ε, θα ανέμενα ε, στην περίπτωση αυτή η ΕΣΜΑ να είναι τμήμα αυτής της συζήτησης που συνεισφέρει με τη δική της εμπειρία. Για παράδειγμα θα ανακύψουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν ε, τη, αφορούν την ισοτιμία των διεθνών υποπτικών ε, ε, συστημάτων και νομίζω ότι εκεί θα συνεισφέρει σημαντικά η ΕΣΜΑ. Επίσης την αποφυγή της ε, διπλής εποπτείας. Η ΕΣΜΑ σίγουρα θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σημαντικό που μιλήσατε λίγο παραπάνω. Εξάλλου είχατε εξοικονομήσει κάποια λεπτά από τις προηγούμενες απαντήσεις σας. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ε, Κάριν Βόρτμαν Κόλ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την ε, υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ιδιαίτερος όταν ε, όσον αφορά την καταπολέμηση υπερβολικών αμοιβών αλλά και ε, υπερβολικών ε, περιουσιακών στοιχείων. Το έχουμε συζητήσει αυτό ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα. Στο Κοινοβούλιο θα θέλαμε να γίνει αυτό για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εσείς θεωρείτε πως οι υποπτικές αρχές θα μπορούσαν να λάβουν μέρος σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Μαγιόρ, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βορτμαρκόλ για την ερώτησή σας. Πιστεύω όντως ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στα μπόνους ε, και την δουλειά που πρέπει να κάνει έσμα. Όλος ιδιαίτερος θα ήθελα να τονίσω τη σχέση ανάμεσα στη ε, μπόνους ε, και τον, την προπτική του καταναλωτή, του μικροεπενδυτή. Ξέρουμε ότι το γεγονός ότι ένας καταναλωτής κατέληξε σε, μια, σε ένα λανθασμένο προϊόν, αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αμοιβέ, αμείβονται αυτοί που δουλεύουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έγινε ολόκληρη συζήτηση για το κατά πόσο οι ενδιάμεση θα πρέπει να πληρώνονται και να κερδίζουν προμήθειες από τους προμηθευτές τους, γιατί εκεί υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον αγοραστή που στο κάτω-κάτω πρέπει να μπορεί να εμπιστευτεί τον σύμβουλό του και να γνωρίζει κατά πόσο οι προμήθειες που κερδίζει ε, παίζουν ρόλο για τις, συμβουλές που του προσφέρει. Ξέρω πως σε πολλές χώρες υπάρχουν σχετικά προγράμματα ώστε να εξασφαλιστεί πως οι προμήθειες ανάμεσα στους συμβούλους ή τους πράκτορες ε, θα εξασφαλιστούν ώστε πραγματικά ο ενδιάμεσος να είναι ανεξάρτητος. Είναι ένα παράδειγμα όπου όντως ένα σύστημα ανταμοιβή έχει αντίκτυπο μεγάλο για τον ε, καταναλωτή και νομίζω πως η ΕΣΜΑ θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στο θέμα αυτό. καθώς και στον ρόλο που παίζουν οι σύμβουλοι διαφόρων ειδών, οι δημοσιολαβητές και ε, μήπως τελικά τα κίνητρα στρεβλώνουν την ε, αγορά. Στρεβλώνουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι σύμβουλοι συμβουλεύουν τους ε, επενδυτές. Uh, thank you very much. And on behalf of the S&D Group, Leonardo Dominici. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ντομένιτσι, σας ευχαριστώ. Το πρόβλημα ε, για το οποίο δημιουργήθηκαν αυτές οι εποπτικές αρχές είναι πάνω απ' όλα η αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου. Εσείς αναφερθήκατε στην αγορά των παραγόγων και η Επιτροπή μας εξετάζει τον κανονισμό που αφορά όντως τα παράγωγα. Το κεντρικό πρόβλημα είναι λοιπόν πώς μπορεί κανείς να έχει τις πληροφορίες, επαρκείς πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ξεπεραστεί αυτή η αδιαφάνεια και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι αυτή της αγοράς. Θεωρείτε πως οι κανόνες που μελετώνται είναι αρκετοί και προβλέπουν τα κατάλληλα μέσα για την ΕΣΜΑ ώστε να μπορεί να έχει τις κατάλληλες πληροφορίες στη διάθεσή της. Πώς ε, πιστεύετε πως θα δοθεί στην ΕΣΜΑ το απαραίτητο κύρος ώστε να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες στη διάθεσή της. I think indeed that the, um, ότι η έλλειψη διαφάνειας στην αγορά των κινητών αξιών ήταν ένας από τους λόγους της νοσιονομικής κρίσης, της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Παραδείγματος χάρη τα credit default swaps. Άμα δούμε τους λογαριασμούς, στο ζενίθ της κρίσης το 8, Ορισμένοι ρυθμιστές χρειάστηκαν, χρειάστηκε να μαντεύουν τους αριθμούς, να τους υπολογίζουν χωρίς να τους έχουν. Δεν είχαν καμία εποπτεία πραγματική για να μπορέσουν να υπολογίσουν επιστημονικά τον κίνδυνο. Νομίζω λοιπόν ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα ως προς την ανάλυση του συστημικού κινδύνου αν υπάρχει επιτήρηση της αγοράς αυτής. Γιατί ο κεντρικός συμψηφισμός δίνει τη δυνατότητα σε μια πιο συνολική εποπτεία και αυτό θα βοηθήσει στην ταύτιση αυτού του συστημικού κινδύνου. Στην περασμένη περίπτωση, στην περασμένη κρίση, αυτά τα credit default swaps ήταν ο κίνδυνος και αν υπήρχε επαρκής επιτήρηση θα είχαν αποφευχθεί. Θα βοηθήσει λοιπόν αυτό βέβαια. Πρέπει να δούμε ποιο μερίδιο της αγοράς θα υπόκειται σε αυτόν τον κεντρικό συμψηφισμό, αλλά φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να υπόκειται. Αναπόφευκτα βέβαια κάποια μερίδια της αγοράς θα ξεφεύγουν, αλλά πρέπει να κατορθώσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο ώστε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς θα την χάνει αυτού του κεντρικού συμψηφισμού. Και όπως είπα και πριν, το πρότυπό μας θα είναι συνδυασμένο σε συνεργασία και με άλλες αρχές καθώς και θα βρίσκεται σε συνεργασία και με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενικά καταρχής που δεν χρειάζεται να τα σχολιάσετε είναι κρίμα νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχει μια παραπάνω γυναίκα εδώ πέρα στις θέσεις που έχουν επιλεγεί. Αναφέρατε αναφέρατε λέγω τα τοξικά προϊόντα και είπατε ότι μερικά θα απαγορεύονται. Ξέρω ότι υπάρχει η δική σας αρχή, αλλά υπάρχουν και οδηγίες που ισχύουν. Είστε απαγορευτής, κυριέ μου. Νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο λύνονται προβλήματα της αγοράς με την απαγόρευση δημοσιονομικών προϊόντων να μας το σχολιάσετε αυτό. Γιατί ξέρω ότι και στην Ολλανδία απαγορεύεται πολλά προϊόντα. Αυτό θα κάνετε και στο Ένωση. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι γυναίκα, αλλά ούτε και απαγορευτής. Προσπάθησα να τονίσω ότι τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή και την καταναλώτρια πρέπει να φτάνουν μέχρι αυτούς μετά από επιλογή, από ελεύθερη επιλογή. Και οι απαγορεύσεις θα είναι κάτι το όλος εξαιρετικό για να τονιστεί ακριβώς αυτό το δικαίωμα της επιλογής και της καινοτομίας. Στη χώρα μου υπήρξαν περιπτώσεις όπου μερικά άτομα δρούσαν στην αγορά, στη χρηματοπιστωτική αγορά, για να έχουν κέρδη χωρίς να βασίζονται καθόλου στις ανάγκες των καταναλωτών και καταναλωτριών. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρξα και εγώ απαγορευτής. Δηλαδή δεν είχαμε δώσει την άδεια χορήγηση τέτοιων προϊόντων. Whatever they would produce, it would be negative for the Γιατί τα αποτελέσματά του ήταν αρνητικά για την αγορά στο γενικότερα, όχι μόνο για τους καταναλωτές και καταναλώτριες, αλλά και για τους προμηθευτές και προμηθεύτριες και θα τα έστρεφε και την φήμη της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τα εξής. Καταρχήν για το short selling. Πρέπει να είμαστε συνεπείς εδώ, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί έχουν αναλυφθεί δράσεις και προγράμματα που δεν συμβιβάζονται με ό,τι έχουν αποφασίσει οι εθνικοί ρυθμιστές. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια λοιπόν. Δεύτερον, ένας ρυθμιστής πρέπει να έχει τη δικαιοδοσία να παρεμβαίνει στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπως το κάνει και για τις κινητές αξίες γενικότερα. Εξαιρετικά βέβαια, όχι κάθε μέρα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία στην πληροφόρηση και αμφιβολία για την ποιότητα της πληροφόρησης αυτής. Σε μερικές περιπτώσεις σταματάει η δραστηριότητα της αγοράς κινητών αξιών επαναλαμβάνω όλος εξαιρετικός και για τα παράγωγα αλλά τελικά πρέπει να σας πω επίσης ότι το short selling καθεαυτό, το design short selling δεν είναι κάτι το αρνητικό. Και γι' αυτό υπάρχουν παραδείγματα. Η περίπτωση Ένρον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί γνωρίζα, ήταν γνωστά τα προβλήματα της εταιρείας αυτής και ήταν γνωστή η περίπτωση να δημιουργήσει φούσκες η δραστηριότητά της. Χρειάζονται λοιπόν και τέτοια μέτρα γιατί καμιά φορά δεν λειτουργούν καλά οι αγορές. Εξαιρετικά το ξαναλέω. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτος γύρος ερωτήσεων για το ΕΛΚ. Κάνει. Πείτε κάνει. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με την καταλληλότητα του πλαίσιο και των εργαλείων, θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη ε, για δύο τα δύο σκέλη. Δηλαδή, ε, η φυστάμενη νομοθεσία σας δίνει αρκετή ε, αρμοδιότητα για να μπορείτε να ενεργήσετε και έπειτα για την μικρο και μάκρο εποπτεία, προληπτική εποπτεία. Πώς αυτή συνδυάζεται με την ε, πρόληψη των συστημικών κινδύνων. Thank you very much. Ε, on current powers. Σας ευχαριστώ πολύ για τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον κανονισμό. Θα ήθελα να πω ότι αρκούν σε αυτό το στάδιο. Έχει πολλή δουλειά μπροστά της η ΕΣΜΑ και πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα αρχίσει η λειτουργία της. Από τη στιγμή που θα αρχίσει κανείς δηλαδή να δουλεύει για, με νέα νομοθεσία, ε, καθώς προχωράει καταλαβαίνει καλύτερα στην πράξη πώς λειτουργεί και επίσης καταλαβαίνει καλύτερα τις αγορές. Για παράδειγμα, αν έχουμε αρμοδιότητες για εποπτεία και θα έχουμε αρμοδιότητες για εποπτεία των ε, CRA, όταν θα αρχίσουμε την αξιολόγηση για την ε, λειτουργία των ΣΥΡΕΙ θα δούμε αν είναι αρκετές οι αρμοδιότητες που έχουμε. Για την ώρα λοιπόν φαίνεται να είναι επαρκείς οι, οι αλλά ε, είναι καινούρια, άγνωστη περιοχή η εποπτεία των CRA. Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχει ξεκινήσει θα δούμε τι λειτουργεί και τι όχι. Και πάντως σίγουρα θα σας ενημερώσω και θα είμαι σαφής όταν δεν πιστεύω ότι είναι ε, επαρκής η αρμοδιότητα. Είναι μια φυσιολογική συνεργασία, αυτό το αναγνωρίζω και από το εθνικό επίπεδο που έχω εργαστεί, όπου κανείς ως ρυθμιστής πρέπει να είναι σαφής ε, για την αποτελεσματικότητα του. Θα πρέπει να πει στους νομοθέτες ας πούμε, ότι χρειάζεται περισσότερη αρμοδιότητες για να είναι πιο αποτελεσματική η εποπτική λειτουργία. Για το συστημικό κίνδυνο, όπως και στην αναρτήριά μου δήλωση, θα συνεργαστούμε στενά με την ΠΥΠΑ και την ΑΙΟΠΑ. Για... νομίζω ότι είχαμε ένα πρώιμο παράδειγμα των αγορών εσύ όπως στο παρελθόν δεν μπορούσαμε να ποπτέψουμε τι συμβαίνει στις κινητές αξίες και αγορές και γι' αυτό και η ΕΣΜΑ πρέπει να μοιραστεί με τους υπόλοιπους επόπτες, τους συναδέλφους, τους κινδύνους που εγκυμονούν σε αυτήν την αγορά. Και επίσης θα πρέπει να συνεργάζεται με το νεόδημητο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Σας ευχαριστώ κύριε Μακάρθη. Θα γνωρίζετε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την ε, έκθεση πρωτοβουλίας για την ε, εμπορία των χρηματοπιστωτικών μέσων για την εμπορία των κινητών αξιών και χρεογράφων. Ιδιαίτερα για την διαφάνεια που αναφέρατε ήδη τρεις φορές στην παρέμβασή σας. Είστε έτοιμος να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες αρχές των ΙΠΑ και να δημοσιεύετε κάποιο μητρό με τους ε, μετόχους ε, της περιλήψης ε, των, των συνεδριάσεων των επιχειρήσεων των ομίλων που είναι γεγραμμένοι στο χρηματιστήριο Ευχαριστώ. Από τα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω, ειδικά με την αναφορήση της Μύφιτ, είναι ότι έχουμε, ότι ένα από τα ωφέλη της Μύφιτ ήταν η αύξηση του ανταγωνισμού ε, νέα ε, και περισσότεροι χώροι, τόποι όπου να γίνονται οι συναλλαγές ε, και νομίζω ότι αυτό ήταν, ήταν μια βελτίωση του περιβάλλοντος και βελτίωση αύξηση του ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα υπήρξε αρνητική επίπτωση μικρότερης διαφάνειας σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών και την ανάκαμψη των τιμών γιατί ορίζονται σε διαφορετικού ε, τόπου συναλλαγή. Άρα λοιπόν υπάρχει το πλεονέκτημα αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων ε, τόπων συναλλαγή. Από την άλλη υπάρχει μεγαλύτερη αδιαφάνεια όσον αφορά τις ε, τιμές και σε κάποιο βαθμό αυτό προσπαθεί κανείς να επιτύχει με την αγορά. Τώρα, υπάρχει ε, μεγαλύτερη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά τις ε, τιμές πριν από τη συναλλαγή και μετά τη συναλλαγή στις διάφορες αγορές. Αυτό είναι ένα από τα θέματα το οποίο θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι της αναθεώρησης MIFID. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί η διαφάνεια εδώ. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της διαφάνειας και του ρόλου των οργανισμών που εποπτεύουμε καθώς και της ε, επιρροής που έχουν, που ασκούν στον ρυθμιστή. Ένα από τα πράγματα που συνηθίζω να λέω στους δικούς μου συνεργάτες είναι ότι αν δεν έχουμε ένα μικρό ταμείο στην ε, πόρτα του οργανισμού και μετράμε πόσοι μπαίνουν μέσα που έρχονται από τις αγορές ε, και πόσοι από την πλευρά των καταναλωτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οργανισμοί τους οποίους επεπτεύομαι ε, είναι καλύτερα οργανωμένοι από τους οργανισμούς στους οποίους εποπτεύουμε. Το ρυθμιστικό ζήτημα θα πρέπει να έχει ψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει ανεξαρτησία από τους οργανισμούς τους οποίους εποπτεύουμε. Και επίσης πρέπει να έχουμε μία ε, ομάδα εκπροσώπησης εντός της ΕΣΜΑ όπου οι συμμετέχοντες στην αγορά να μπορούν να συμμερίζονται, να ανταλλάσσουν υπόψη με τον ρυθμιστή υπάρχει ε, διαφάνεια ε, σε σχέση με αυτό το τύπο άσκησης ε, επιρροής, σε σχέση με την εξέλιξη διαβουλεύσεων. Νομίζω ότι χάρη της... Νομίζω ότι το επίπεδο των λεπτομερών των λεπτομεριών θα είναι επαρκώς ρυθμισμένο ώστε να εξασφαλίσει τη δική μας αυτονομία. Θα δημοσιεύεται ε, πληροφορίες είναι η ερώτηση. Ναι, θα δημοσιεύονται ε, πληροφορίες εκ μέρους των συμμετεχόντων στην αγορά. Ναι, ήταν πολύ ειδική η ερώτησή μου. Πολύ συγκεκριμένη. Σε σχέση με... Ναι, θα δημοσιεύουν, θα κοινοποιούνται οι πληροφορίες για τις συναντήσεις με συμμετέχοντες της αγοράς. Πρόεδρος, ωραία λοιπόν έχει ολοκληρωθεί. Ε, ξεκινάει ο τέταρτος γύρος. Ε, ε, βάσει του ρολογιού μπορούμε να επιτρέψουμε ακόμα λίγες ερωτήσεις. Θα είμαι πολύ αυστηρή σχέση με τήρηση της σειράς αγόρευσης των εκπροσώπων των ομάδων. Ο Πίτερ Σκίνερ, συνεπώς, έχει πρώτος το λόγο. και Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, ε, αναφερθήκατε στην ε, αποτελεσμότητα του προηγούμενου συμβουλίου της ΕΣΜΑ και είπατε ότι είχε μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Ποια ε, ήταν τα πλεονεκτήματα ωστόσο και πώς ε, φαντάζεστε εσείς μια περαιτέρω διεύρυνση των δικών σας αρμοδιοτήτων στο μέλλον. Αναφερθήκατε επίσης στο ζήτημα των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Σε ποιο βαθμό θα αναλάβουν οι οίκοι αυτοί μια ευθύνη για τις αποφάσεις τους. Το, τέλος, το σημαντικότερο θέμα της αξιολόγησης ε, του δημόσιου χρέους τι προβλέπετε, ποιο χρονικό διάστημα προβλέπετε για την επίλυση του ζητήματος του δημόσιου χρέους. Τέταρτον, οι εποπτικές αρχές θα έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν ορισμένα προϊόντα υψηλού κινδύνου για μια συγκεκριμένη περίοδο. Ποια είναι η εμπειρία που είχατε μέχρι τώρα και ποια είναι η αναλογία των απαγορευμένων προϊόντων. Είπα στην αρχή ότι θα πρέπει να περιορίζετε το χρόνο ομιλία σας. Παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας τέθηκαν. Θα έλεγα ότι ήταν δύσκολο να κατανοήσω τη μετάφραση. Ίσως δεν ε, κατάλαβα πλήρως τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, δεν ε, έχω συνομιλήσει με τους εκπροσώπους τους σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ε, έχω εμπειρία βεβαίως στην, ε, στον τομέα του ελέγχου και υπάρχουν κάποιες ομοιότητες αλλά και διαφορές. Οι CRAs παρέχουν κάποιες ε, διασφαλίσεις για τους κινητούς τίτλους Εξετάζοντας λοιπόν τις παρούσες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους CRAs, ε, πιστεύω θα υπάρχει σημαντικός, ε, σημαντική αποτελεσματική χρηματοπιστωτική εποπτεία. Όσον αφορά τώρα τη μείωση του ελλείμματος, δεν νομίζω ότι αυτό υπάγεται στα όρια της αρμοδιότητας της ΕΣΜΑ. Το δημόσιο χρέος αφορά τις αντίστοιχες χώρες που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μειώσουν τα χρέη τους. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι εμπίπτει το θέμα αυτό στην αρμοδιότητα της ΕΣΜΑ. Ο Πίτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ε πώς βλέπετε το ρόλο της κοινή επιτροπής και ποιε είναι οι δικέ σα φιλοδοξίε σε σχέση με την συνεργασία με την ε, Μικτή Επιτροπή. Απάντηση. Περιμένω να υπάρχει ιδιαίτερο ανεργή συνεργασία με την ΙΜΠΑ και την ΑΙΟΠΑ, γιατί όλοι αυτοί οι οργανισμοί ασκούν την ε, ε, χρηματοπιστωτική υποπτία και βεβαίω αυτό είναι σε αποχρόν λόγο συνεργασία. Ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η χρηματοπιστωτική όμιλη, όπου και οι δύο παρέχουν ασφαλίσεις, τραπεζικές ε, υπηρεσίες κλπ. Και εδώ είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα που θα υπάρξει συνεργασία, γιατί αλλιώ δεν είναι δυνατόν να είναι κανεί αποτελεσματικό ω ρυθμιστή. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά επίση την πλευρά των καταναλωτών, των επενδυτών στον τομέα τη λιανική. Υπάρχουν ορισμένα προϊόντα όπου υπάρχει ένα στοιχείο ασφάλεια σε συνδυασμό με ένα στοιχείο επένδυση ή ένα στοιχείο επάνδυση, ε, συνδυασμένο με ένα στοιχείο τραπεζικό. Εάν θέλετε λοιπόν να δουλέψετε με αυτά τα προϊόντα, ε, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους δύο άλλους ρυθμιστές στον τομέα της ασφάλισης και της, ε, των τραπεζών, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα αυτών των προϊόντων. Και σε ακραίε περιπτώσεις θα πρέπει να προσέξει κανεί τις τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία με την αρχή ασφαλίσεων και την ε, αρχή τραπεζών. Ένα τελευταίο ερώτημα, ο Πασκάλ. Ευχαριστώ. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που αναλάβατε ενώπιον μας τη δέσμευση να κοινοποιείτε τα πρακτικά των συναντήσεων με τους συμμετέχοντες που προέρχονται από την ε, χρηματοπιστωτική βιομηχανία και βεβαίως θα είμαστε ιδιαίτερες ε, προσεκτικοί όσον αφορά αυτή την ε, εφαρμογή, την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης που αναλάβατε. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο κρίνετε ότι έχετε ως ρυθμιστής επαρκείς πληροφορίες για να υλοποιήσετε την οδηγία για, την κατάχρηση, για το market abuse και να μας πείτε κατά πόσο ορισμένοι παίκτες της ε, αγοράς προσπαθούν να χειραγωγήσουν τις αγορές ε, μέσω των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών, των egg sellings. Για παράδειγμα, αυτό γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και όπου εκεί επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο επίση συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια είναι η δική σα θέση επί τούτου. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία όσον αφορά την ε, κατάχρηση της αγοράς. Um, Και πάλι θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση με την αγορά χρεογράφων όπου οι ρυθμιστές έχουν την ε, δυνατότητα να σταματήσουν τις συναλλαγές αλλά και να ενεργήσουν κατά της χειραγώγησης από διάφορους φορείς της αγοράς και μάλιστα πρόσφατα στο δικό μου οργανισμό είδαμε ένα μέρος που όντως προσπαθούσε με μικρές συναλλαγές στο τέλος της ημέρας να, να επηρεάσει την, την τιμή της συγκεκριμένης μετοχής. Ναι, πρέπει να, να έχουμε αρμοδιότητες ώστε να ενεργήσουμε σε περίπτωση χειραγώγησης όχι μόνο για τις αγορές χρεογράφων αλλά και για τις νέες αγορές που θα εποπτεύσουμε για το κατά πόσο τώρα το short selling ήταν πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής είναι μανάμεκτες Και ως αποτέλεσμα αυτού του νέου ρόλου στις αγορές ΟΗΣΗ θα έχουμε μεν καλύτερη εικόνα των αγορών, αλλά έχουμε επίσης συμφωνήσει πως ορισμένα από αυτά τα προβλήματα με τα χρέη, τα κρατικά, σχετίζονται με θεμελιώδη ζητήματα στην οικονομία της χώρας. Ε, τώρα, το, να δούμε σε ποιο βαθμό υπήρξε χειραγώγηση δεν ξέρουμε. Ακούμε διάφορες ιστορίες από διάφορους ρυθμιστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι νέοι κανόνες θα μας δώσουν καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, αλλά εν γέννη θα πρέπει να έχουμε την ερμοδιότητα αυτή, όπως και στις αγορές χειρογράφων εάν υπάρχει χειραγώγηση, να μπορούμε να ενεργήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ τέλος ε, της ακρόασης. Καταφέρατε να είστε σύντομος και να μείνετε μέσα στα χρονικά όρια. Ε, και μπορέσαμε να ακούσουμε δύο επιπλέον ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να αποχωρήσετε τις αιθούσεις. And we have another hearing, so don't leave. Φύγετε, έχουμε άλλη ακρόαση. Right. Everybody, Παρακαλώ. Υπάρχουν θέσεις πίσω. Τώρα περνάμε στη δεύτερη μας ακρόαση του Γαβριήλ Μπερναρντίνο που έχει επιλεγεί από τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Για την περίπτωση που έχουν έρθει μερικοί τώρα θα σας υπενθυμίσω ότι στην αρχή θα κάνει μία εισαγωγή πεντάλεπτη ο άνθρωπος και μετά θα γίνουν ερωτήσεις και διάλογος. Ένα λεπτό για τις ερωτήσεις και τρισήμιση λεπτά για την απάντηση, για τις απαντήσεις. Σας ξαναλέω, μην θέσετε πολλαπλές ερωτήσεις. Αν συνδέονται βέβαια δύο εντάξει, αλλά τρεις και πάνω νομίζω ότι θα σας θέσω εκτός θέματος. Παρακαλώ λοιπόν μην το κάνετε, είναι άχρηστο και άδικο. Λοιπόν, ο Γαβριήλ για την εισαγωγή του. Χα, χα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, μέλη της Επιτροπής οικονομικών και νομισματικών θεμάτων. Πιστέψτε με, είναι μεγάλη χαρά η παρουσία μου εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να σας παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις για την αρχή της εποπτείας που, της οποίας προεδρεύω. Ζούμε δύσκολη περίοδο χρηματοπιστωτική κρίση έχει αμφισβητήσει τη δυνατότητα οποιοδήποτε επόπτη να αντεπεξέλθει. Και πιστεύω ότι αυτό απαιτεί δράση και όραμα. Ο καθορισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων δίνει μια ευκαιρία να υπάρξει επιτέλους αυτή η εποπτεία πράγμα το οποίο θα ωφελήσει πολύ στο στόχο προς την, της ε, σταθερότητας και θα ωφελήσει επίσης τους καταναλωτές, καταναλώτριες και την βιομηχανία. Κάτε με, η ΕΑΕΣ πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα για να το κατα, τα καταφέρει. Πρώτον, την ανεξαρτησία της. Κάτε με, η ανεξαρτησία πρέπει να φαίνεται από τις πράξεις μας, από τη χρήση των δικαιοδοσιών μας, εάν είμαστε αδέκαστοι και συνεπείς. ανεξάρτητοι από τους ενδιαφερόμενους, από τη βιομηχανία, από την Κομισιόν και από τα ίδια τα μέλη. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να υπάρχουν ήδη οι πόροι μας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει η ΕΑΕΣ να μπορεί να χρησιμοποιεί την ε, γνώση που διαθέτουν τα μέλη της. Επίσης πρέπει να εφαρμόσει ένα σωστό σύστημα διαχείρισης με βάση τις αρχές της διαβούλευσης, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας και πρέπει να εκμεταλλευτεί την εμπειρία των διαφόρων επιτροπών ενδιαφερομένων. Ε, μαζί με την καλή διαχείριση υπάρχει βέβαια και η ανάγκη να, υπάρχει, να δίνονται, να είναι υπόλογοι οι ΕΑΕΣ στα μέλη της και σε εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρέπει να είναι έτοιμη και πρόθυμη να συζητήσει και να κάνει ανταλλαγές απόψεων ανα πάσα στιγμή. Η ΕΑΕΣ είναι δίκτυο εποπτών αλλά πρέπει να αποδείξει ότι είναι χρήσιμη, χρησιμοποιώντας πρωτοβουλίες εκπαίδευσης εποπτών, ας πούμε, και μέσω της διαχείρισης μιας κεντρικής τράπεζας δεδομένων για να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης και καθορισμού χρήσιμων δικτών. Ταυτόχρονα αυτό δεν είναι απλή συνέχιση προηγούμενης εθνικής εμπειρίας. Είναι και κάτι το καινούριο, θα έχει και καθαρά δικές της δικαιοδοσίες κατά την εποπτεία, την προετοιμασία δοκιμών, την διευθέτηση διαφορών και την εφαρμογή προστασίας καταναλωτών και καταναλωτριών και πρέπει να συνεργάζεται με τις άλλες εποπτικές αρχές μέσω της Μικτής Επιτροπής και θα συμβάλλει στην γενικότερη αξιολόγηση που θα γίνεται τακτικά. Για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει η ΕΑΕΣ να έχει γνώση, εμπειρία και ηγεσία. Αυτές είναι μερικές από τις αξίες που ταπεινά μπορώ να σας χορηγήσω. Κατά τη σταδιοδρομία μου στην εποπτεία και στις ασφαλίσεις και στις συντάξεις εθνικά και διεθνώς Έχω πιστεί για την αξία του διαλόγου, αλλά και για την ανάγκη να είμαστε αποτελεσματικοί. Έχω νομίζω το σωστό όραμα για να ηγηθώ της ΕΑΕΣ και να πετύχω τους στόχους της. Είμαι υπεύθυνο και ενεργός και ανεξάρτητος. Πιστεύω πραγματικά στο ευρωπαϊκό όραμα. Τέλος με μεγάλο πάθος πραγματοποιώ την εργασία μου, δεν μπορώ να την πραγματοποιήσω αλλιώς. Διότι πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα είναι σημαντικά, αλλά οι άνθρωποι τελικά κάνουν τη διαφορά. Και ελπίζω ότι με την ε, υποστήριξή σας θα πετύχει η ΕΑΕΣ και φυσικά είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε τυχόν απορίες. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Αρχίζουν οι ερωτήσεις ο πρώτος γύρος εξ του ΕΛΚ ο Ζαν Πολ Γκαβζής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Βερναρδίνο. Θα θέσω το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον προηγούμενο και θα θέσω και στον επόμενο. Είπατε στο τέλος ότι οι άνθρωποι μετράνε. Πράγματι. Αυτό που μας ενδιαφέρει και μας ανησυχεί μας είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι διορισμοί, οι θέσεις σας στην ιεραρχία και ορισμένοι αναρωτιόμαστε μήπως οι επιλεγέντες δεν έχουν όλη την απαραίτητη δικαιοδοσία που χρειάζονται και ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα που έθεσε μεταξύ άλλων και το Κοινοβούλιο. Σας ερωτώ λοιπόν κύριε Βερναρδίνο, πώς θα καταφέρετε από τη θέση που έχετε τώρα να περάσετε στην αυριανή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκοζέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κατανοώ το ερώτημά σου, κατανοώ. Και για μένα είναι μεγάλη τιμή που επελέγει από τους ομολόγους μου ως πρόεδρος. Νομίζω ότι έχω και την εμπειρία και την αρχαιότητα. Το έχω αποδείξει ότι είμαι σε θέση να ηγηθώ συλλογικών σωμάτων και το έχω πράξει και διεθνώς προεδρεύοντας σε ομάδες εργασίας, σε περιπτώσεις πτωχεύσεων Έχω κάνει συζητήσεις με το Συμβούλιο για πτωχεύσεις. Εργάστηκα με τους συναδέλφους μου σε, διάφορες, σε διάφορες εποπτικές αρχές και έχω νομίζω και την αναγνώριση τους. Καταλαβαίνω βέβαια ότι θα πρόκειται για κάτι το καινούριο, δηλαδή για μια διαδικασία όπου δεν πρόκειται όπως το παρελθόν να, να ζητούμε πάση θυσία συνένεση, την επίτευξη πάση θυσία συνένεσης. Αλλά θα βασιζόμαστε στις βέλτιστες πρακτικές. Μέσα στα πλαίσια βέβαια του ισχύοντος κανονισμού, βάσει του οποίου ο πρόεδρος πρέπει να έχει το όραμά του εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εποπτών, αλλά έχω τις απόψεις μου και πρέπει νομίζω η Προεδρία να έχει απόψεις. Οι δε απόψεις μου νομίζω ότι γίνονται σεβαστές από τους υπόλοιπους. Με βάση το λέω αυτό την εμπειρία μου. Πιστεύω πραγματικά ότι για να μπορέσει η ΕΑΕΣ να πετύχει χρειαζόμαστε κάποιον που να μπορεί να μιλάει την ίδια γλώσσα με τους υπόλοιπους επόπτες. Να καταλαβαίνει ποιες είναι οι διαφορές, αλλά ταυτόχρονα να έχει και, μία, και ένα σαφές όραμα για το μέλλον και για την πρόοδο. Και νομίζω ότι το όραμα αυτό το έχω. Άρα πληρώ τους όρους νομίζω για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου κύριε Γκοζέση. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερο ερώτημα. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών ο Πέτρος Σκίνερ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Μπερναντίνο, Πρόεδρος φυσικά, αν περάσετε αυτήν την ακρόαση δηλαδή, θα είστε ένας πολιτικός ηγέτης για τις χρηματοπιστωτικές αρχές είπατε ότι θα καταδιηγηθείτε από τις καλύτερε πρακτικέ. Αυτό είναι το όραμά σας. Πώς θα το κάνετε αυτό στο πλαίσιο της, κοινή, της Μικτής Επιτροπής, που είναι ένα κενό κουτί στην ουσία αυτή τη στιγμή στην ε, νομοθεσία που έχουμε συντάξει. Θεωρείτε πως είναι μια φιλόδοξη τρύπα που πρέπει να πληρωθεί, ένα και χάσμα που πρέπει να πληρωθεί από τα στάνταρ και τις πρακτικές των τριών ε, ε, οργανισμών, των τριών αρχών. Ευχαριστώ πολύ Πίτερ για αυτή την ερώτηση. Πιστεύω πως η Μεκτή Επιτροπή είναι ένα σημαντικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας Νομίζω πως πρέπει να οικοδομήσουμε σε μια προσέγγιση βήμα προς βήμα αυτή τη διαδικασία της συνεργασίας. Έχουμε κάποια εμπειρία από το παρελθόν. Αν με ρωτήσετε εμένα, το παρελθόν είναι μια καλή αναφορά στις θέματα συνεργασίας και νομίζω πως ε, σε ορισμένες περιπτώσεις όχι τόσο καλή αναφορά. Αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλους τομείς όπου οι τρεις αρχές ε, να συνεργάζονται. Θα πρέπει να δεσμεύσουμε πόρους στους τομείς αυτής για τα χρηματοπιστωτικά κούσο μήλους για παράδειγμα για την προστασία του καταναλωτή φυσικά εκεί θα πρέπει να ε, οικοδομήσουμε συνεργασίες. Υπάρχουν πολλοί τομείς όπου δεν θα πρέπει να υπάρχει χώρος για διαφορετικές απαντήσεις και όπου φυσικά χρειάζεται να συνεργαστούμε. Εγώ θα είμαι μια φωνή στην κοινή επιτροπή. Θα είμαι βέβαια η φωνή των ασφαλίσεων και των συνταξιδοτικών ταμείων. Αλλά σίγουρα θέλω να βελτιωθεί για το μέλλον αυτή η συνεργασία. Φυσικά το να εργάζεται κανεί στη Μικτή Επιτροπή δεν σημαίνει πω θα καταλήξει σε ενιαίες λύσεις στα διάφορα προβλήματα. Πιστεύω πως οι ασφαλίσει και οι συντάξει, οι ρυθμίσεις και η εποπτεία θα μπορούσαν να φέρουν θέμενη αξία. Δεν πρέπει πάντοτε να υιοθετούμε τραπεζικέ συστήματα ε, και λύσεις. Πρέπει να μάθουμε από με αυτό το πνεύμα θα μπω στην Κοιμικτή Επιτροπή, θα προσπαθήσω να δημιουργήσω πρόοδο, αλλά και να σεβαστώ τις διαφορές εκεί που υπάρχουν. Thank you very much. Uh, and now... Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος της Άλντε, ο Όλη Σμιτ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το ίδιο θέμα όπως ο Πίτερ Σκίνερ γιατί πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό. Όπως ίσως γνωρίζετε η φιλελεύθερη ήθελε μία αρχή γιατί δεν θα λέγαμε πως η δική σας αποστολή ας πούμε δεν ε, χρειάζεται να υπάρχει, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ακόμα και αν στην κοινή επιτροπή θα μπορούσατε να καλύψετε πολλά κενά, πιστεύουμε πως υπάρχουν προβλήματα. Εσείς θα προσπαθήσετε να κάνετε κάποια βήματα ώστε να ενσωματωθούν οι τρεις αρχές να συνεργαστούν με βαθύτερο τρόπο. Θα μπορούσε αυτό να αποτελεί φιλοδοξία για σας ως πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σμιτ. Γνωρίζω βεβαίως ότι η θέση σας είναι ιδιαίτερα δρυμία σε αυτό το τομέα, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη μου είναι μια σταδιακή προσέγγιση. Για την ε, ώρα νομίζουμε, πιστεύω πως είναι σωστή η λύση των τριών διαφορετικών αρχών, να υπάρχει δηλαδή διάκριση. Στο μέλλον, στα επόμενα δύο-τρία χρόνια και φυσικά ο κανονισμός προβλέπει τέτοιου είδους ανάλυση στο μέλλον, ε, θα δούμε λοιπόν πού κατευθύνονται οι αγορές γιατί πιστεύω πραγματικά πως υπάρχουν τομείς όπου χρειάζεται να συνεργαστούμε, να δώσουμε νέες απαντήσεις. Όμως δεν θα πρέπει, όπως σας είπα και απαντώντας στον ε, Πίτερ, ότι θα πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό ήταν λάθος στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και να μάθουμε. Εμένα πως Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι εγώ θα συνεργαστώ μαζί με τους συναδέλφους ώστε να φτιάξουμε μια ισχυρή δέσμευση όπου αναπτύσσονται οι διατομεακοί κίνδυνοι. Να μην υπάρχει δηλαδή δυνατότητα όπως στο παρελθόν η μεταφορά ε, των, να μεταφερθούν μάλλον οι κίνδυνοι, να έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε ε, κάθε φορά από μία σκοπιά. Εγώ θα είμαι ανοιχτός ε, απέναντί σας. Ένας από τους φόβους μου για μια απόλυτα ενωπημένη αρχή είναι το γεγονός πως ε, ε, ως συνήθως και το έχουμε δει ήδη σε κάποιες χώρες ο τραπεζικός τομέας και εύλογα είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα. Όμως σε μια κατάσταση όπου, όπου είμαστε, όπως αυτή που είμαστε τώρα με την εφαρμογή της Solvency 2 που θα εφαρμοστεί το 2013 θα χρειάζεται να έχουμε δικαιωμένους ανθρώπους και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες. προτεραιότητες όπου αν έχουμε μια ευ... είχαμε δηλαδή μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή δεν θα μπορούσαμε να τις ιεραρχήσουμε σωστά. Χρειάζεται χρόνος λοιπόν για να, να, να δρομολογηθούν όλα αυτά. Δεν θέλω εγώ από, να δουλεύω σε αποκλεισμό ή μόνος μου. Όχι, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όμως η αγορά, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και όλα το καθεξής και όλα αυτά να αξιολογηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εκ μέρου των Πρασίνων ο Σφεν Γκίγκολτ έχει το λόγο. Ναι, ε, γεια σας. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σε σχέση με την αρκτήρια ομιλία σας. Αναφέρεται ε, τα μέλη των εποπτικών ρυθμίσεων ως ε, πελάτες. Really not Uh, Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό δεν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε το πνεύμα του θεσμικού εργάνου. Ε, αναφερθείτε επίση σε ένα δίκτυο. Ε, δεν πρόκειται για ένα δίκτυο και δεν είναι τα μέλη επόπτες που είναι οι πελάτες σας. Είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είστε υπόλογος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για μας αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά τώρα, για να έρθω στο ερώτημά μου. Θα ήθελα να μας πείτε πώς, χρησιμοποιείτε, πώς θα χρησιμοποιήσετε τις εξουσίες σας ούτως ώστε να επεξεργαστείτε μια αυστηρότερη ρύθμιση για τους ε, ε, συστημικούς οργανισμούς στον τομέα της ασφάλισης. Ε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις χρηματοδότησης που θα θεσπίσετε για αυτά τα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη, γιατί μια ενδεχόμενη αποτυχία θα, είναι εις βάρος των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γκίγκολ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σχολιάσω στα όσα είπατε για την, τα εισαγωγικά μου λόγια. Νομίζω ότι ε, πράγματι οι, όλες οι εποπτικές αρχές συνιστούν ένα δίκτυο εποπτείας. Βεβαίως ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατατείνουμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό κοινό αγαθό που είναι το ευρωπαϊκό κοινό συμφέρον, αλλά υποφάσεις στο επίπεδο της ΕΑΕΣ θα λαμβάνονται από τους Ευρωπαίους ε, ρυθμιστές. Όταν είπε ότι η ΕΑΕΣ μπορεί να επιφέρει προσθέμενη αξία για τα μέλη της, αυτό το είπα υπό την έννοια ότι μία από τις εξουσίες της ΕΑΕΣ, για παράδειγμα, θα είναι να ε, διερευνά ενδεχόμενε παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Νόμου. Βεβαίως, εάν μπορείτε ταυτόχρονα να το κάνετε εκ των προτέρων, ούτως ώστε να έχετε επαφές με τις εποπτικές αρχές για να μπορέσετε να προλάβετε ε, μελλοντικέ εσφαλμένες εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Νόμου, νομίζω ότι αυτή είναι μια προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τα μέλη μας, όχι να λειτουργήσουμε ενάντια στα μέλη μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα ε, των ρυθμιστικών αρχών. Ένα από του σημαντικού τομεί που αναφέρεται είναι ο τρόπο που θα προσεγγίσουμε το συστημικό κίνδυνο. Και όπω ξέρετε γίνεται τεράστια συζήτηση σε σχέση με το συστημικό κίνδυνο και τι ασφάλειε. Ε, κάτι που είναι σίγουρο είναι ότι ο κίνδυνο τη ασφάλεια διαφέρει από το συστημικό κίνδυνο στο μέτρο των τραπεζών, λόγω ακριβώ τη ε, φύση αυτή τη δραστηριότητα που είναι εντελώ διαφορετική. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ασφάλειες και συντάξεις βεβαίως δεν μπορούν να ενέχουν συστημικά προβλήματα, συστημικούς κινδύνους για τις αγορές. Βεβαίως μπορούν να διευρυνθούν εάν υπάρχει συστημικός κίνδυνος από τον τομέα των τραπεζών. Ε, για παράδειγμα χρησιμοποιούν ε, οι ασφάλειες θεσμικούς επενδυτές ε, και οι συντάξεις και η δραστηριότητα του τομέα αυτού αντανακλά, των τραπεζών τραπεζικού τομέα, αντανακλά βεβαίως τον κλάδο των ασφαλίσεων και των συντάξεων. Και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για να αναγνωρίσουμε κάποιους δείκτες για την καταμέτρηση, την αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου και η προσπάθεια αυτή θα γίνει και από την πλευρά των τραπεζών. Τώρα, ποια εργαλεία έχουμε για να προλάβουμε αυτού του συστημικού κινδύνου. Επιτρέψτε να σας πω ότι πιστεύω πραγματικά στο ρόλο της εποπτείας και θα ήταν περίεργο εάν ε, δεν το πίστευα. Και βεβαίω ε, θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση που να βασίζεται στο συστημικό κίνδυνο στο επίπεδο τη πρόληψη, τη πρόβλεψη. Και ε, βεβαίως ε, οι θεσμικοί οργανισμοί θα πρέπει να προσελκύουν περισσότερη εποπτεία, να υπάρχει περισσότερη παρεμβατική εποπτεία και μεγαλύτερη συγκέντρωση πληροφοριών. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εποπτεία χωρίς να βασίζεται σε πληροφορίες αλλά επίσης να υπάρχουν ε, κεφαλακές απαιτήσεις, κεφαλακή επάρκεια που να βασίζεται σε συστημικούς κινδύνους, στην εκτίμηση συστημικών κινδύνων. Όμιλοι που ε, ενέχουν περισσότερους κινδύνους θα προσελκύσουν περισσότερα κεφάλαια και αυτό εξορισμό Ε, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό σε όλη αυτή τη συζήτηση σε σχέση με συστημικό κίνδυνο κλπ. Ας δούμε την ε, σωρευτική επίδραση. Ε, δεν θα έπρεπε νομίζω απλώς να θέτουμε απαιτήσει επί απαιτήσεων χωρίς να εξετάζουμε το σωρευτικό αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι με το Solvency 2 έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας ασφαλιών ε, που θα έχουν ε, κεφαλική επάρκεια για να αντιμετωπίσουν το συστημικό κίνδυνο που θέτουν. Ευχαριστώ. Ε, για τι συντάξει. την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή ψήφισε μια έκθεση για τι συντάξει και επισημάναμε ότι οι συντάξει θα πρέπει να δέπτουν σε αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών μελών. Επίση, τονίσαμε την ανάγκη οι χώρε μέλη να εφαρμόσουν την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και να βελτιώσουν τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για την ε, μεταφορά συντάξεων από χώρα σε χώρα. Τώρα, όσο αφορά την οδηγία, ε, έχω κάποια ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί σε ορισμένε χώρε. εσείς ε, ως πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος, ε, θα έχετε την εξουσία να αναφέρετε στις ε, εθνικές αρχές ότι δεν εφαρμόζεται επακριβώς αυστηρά η νομοθεσία στο επίπεδο χωρών. Πώς θα ασκήσετε αυτό το ρόλο σας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία Φόρντ. Οι ευρωπαϊκές συντάξει είναι πολύ σημαντικό θέμα πολλές φορές θεωρούνται αρνητικές διότι οι ασφαλίσεις μας ενδιαφέρουν περισσότερο αλλά εγώ δίνω την ίδια σημασία και στις συντάξεις. Έχω εργαστεί επί των συντάξεων πολλά χρόνια και μου αρέσει αυτό το θέμα, μου αρέσουν οι συντάξεις. Κατανοώ βέβαια ότι πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας για τις συντάξεις. Και βέβαια η και η ίδια η οδηγία είναι οδηγία με εναρμόνισης. Ανάλογα με τον τομέα βέβαια. Αλλά όπως είπατε και εσείς η ΕΑΕΣ θα έχει τη δικαιοδοσία να κάνει αναλύσεις και κρίσεις για την εφαρμογή αυτών που θα προβλέπουν τα κράτη-μέλη και είναι ζωτικό να έχουμε προσωπικό που να καταλαβαίνει τι γίνεται με τις συντάξεις που διαφέρουν από τις τράπεζες και τις ασφαλίσεις. Έχει ιδιαιτερότητες οι συντάξεις. Και εγώ νομίζω ότι είμαι σε θέση να κάνω τέτοιες αναλύσεις γιατί έχω εμπειρία στην εφαρμογή διατάξεων και για τις ασφαλίσεις και για τις συντάξεις και εθνικά και ενωσιακά. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να αναφέρω λίγο το όραμά μου για τις μελλοντικέ συντάξεις. Όλοι αναγνωρίζουμε σήμερα τη σημασία που έχει ο δε, που οι συντάξεις δευτέρου και τρίτου πυλώνα στις αγορές. Και φαντάζομαι ότι αναρωτιέστε κι εσείς πώς συνδέονται οι συντάξεις με τις πιτοχεύσεις. Εγώ είμαι διαφανέστατος. Ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλοι για αυτό το θέμα. Υπάρχει χώρος βελτίωσης στη διευθέτηση των συντάξεων στην Ευρώπη. Σε πολλούς τομείς μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, όπως τη διαχείριση των ίδιων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και σχημάτων ή σε θέματα ασφαλείας των συντάξεων και ελπίζω να μπορέσω να συμβάλλω και σε αυτό. Βέβαια δική σας δουλειά είναι και της Κομισιόν τελικά, καθώς και του Συμβουλίου, αλλά εγώ ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω τα τρία αυτά όργανα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος για το ΕΛΚ, ο κύριος Νίτρας. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετίζω διότι φαίνεται ότι η προσωπική σας, ότι οι ικανότητές σας και η εμπειρία σας είναι μια εγγύηση για μας. Μιλήσατε για συντονισμό δικτύων άλλων εποπτικών οργανισμών που έχουν και αυτοί τις δικαιοδοσίες τους. Ερωτώ λοιπόν, σε τι βαθμό είστε πρόθυμος και διατεθειμένος, σε τι βαθμό βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα για σταθεροποίηση των τοπικών αγορών, ιδιαίτερα μετά το νέο σύστημα υπολογισμών που θέτει και νέα κριτήρια. Γιατί υπάρχει ο φόβος οι εποπτικές αρχές, οι εποπτικές λέω αρχές λέω, να βρεθούν σε μια θέση όπου θα αποσταθεροποιούν τις τοπικές αγορές. Και επομένως εδώ φαίνεται η σημασία της πανενοσιακής εποπτείας. Τι φρονείτε κι εσείς επ' αυτού. Ευχαριστώ κύριε Νίτρα. Ο ρόλος της ΕΑΕΣ, συντονισμού δηλαδή και δράση στα μέλη της είναι ζωτικός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσει και προβλήματα για τους εθνικούς επόπτες. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δικαιοδοσιών. Η καθημερινή εποπτεία είναι τοπική. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα ασχολούνται με το συντονισμό των δραστηριοτήτων των τοπικών εποπτών. Και βέβαια θα είναι υπεύθυνε για την παρακολούθηση του κατά πόσον γίνονται σωστά οι εποπτείες και αυτά που προβλέπει ο νόμος. Ως προς δε, τις τα νέα κριτήρια που αναφέρατε για τις ασφαλίσεις, τρία πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Να υπάρξει εξισορροπημένη προσέγγιση φρόνιμη. Δεύτερον, είναι επίσης σημαντικό να δούμε ποια ακριβώς είναι η δυσκολία του πράγματος, πράγμα που δεν σημαίνει ότι χρειάζονται δύο χωριστά συστήματα για τις μεγάλες και για τις μικρές χώρες. Ένα σύστημα, αλλά με τις απαραίτητες απλοποιήσεις και προσαρμογές για τη χρήση του. ώστε να μπορούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να δρουν στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μας και από αυτού θα επιμείνω. Τρίτον, κάτι το οποίο ήδη αρχίζει να εφαρμόζεται, να υπάρξουν σωστές μεταβατικές περίοδοι, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τις μικρότερες χώρες και επιχειρήσεις καθώς και με μονομένους επόπτες και επόπτριες. Να υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι για την προσαρμογή του συστήματος στο αφορά τις πιτοχεύσεις χωρίς διακοπή η ρήξη. Και δεν νομίζω ότι η ΕΑΕΣ θα παίξει ασήμαντο ρόλο εδώ. Αντίθετα, πιστεύω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κοινό πλαίσιο εποπτείας στην Ευρώπη. Γιατί αυτό θα δείξει πόσο χρήσιμο είναι, από μόνο του θα φανεί. Στα χρηματοπιστωτικά συστήματα ιδιαίτερα θα πρόκειται για το πρώτο τέτοιο πλαίσιο εποπτείας. Άλλο είναι να υπάρχουν οδηγίες και κανονισμοί και άλλο η εφαρμογή του στην πράξη. Ένα κοινό πλαίσιο εποπτείας είναι κάτι πολύ χρήσιμο για το μέλλον. Θα είναι. Και αυτό είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσω. Και τώρα για τους σοσιαλιστές, κυρία Φέιρο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και είναι μεγάλη χαρά μας που βρίσκεται εδώ μεταξύ μας. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξή. Αληθεύει ότι όποιος ε, πρώτος ε, αναλαμβάνει μια θέση έχει με μεγάλη ευκαιρία να δώσει μορφή και να σημαδέψει, να καθορίσει τις γραμμές ε, της μελλοντικής του δράσης. τώρα, η ο τομέας αυτός ε, θα δει πολλές εντάσεις λόγω της γύρανσης του πληθυσμού αλλά και λόγω των θεμάτων ε, εθνικού χαρακτήρα ε, που δεν υπάρχουν σε σχέση με τις υπόλοιπε εταιρείε. Στην άσκηση λοιπόν της δικής σας εντολής τι ρόλο θα παίξετε όσον αφορά την υπεράσπιση του καταναλωτή και του πολίτη, των δικαιωμάτων του πολίτου σε σχέση με τις ε, επαγγελματικέ συντάξεις. Θα είναι κρίσιμη η θέση σας. Ε, ποια θα είναι η πιο σημαντική σας ε, λειτουργία, η ενίσχυση της νομικής βάσης επί της οποίας θα λειτουργήσετε στη θέση αυτή ή η υπεράσπιση της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα αγγλικά. I think that it's... Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι δηλαδή όποιος πρώτος ε, καλύψει μια θέση, νεόδυνη θέση, θα έχει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό της μελλοντική λειτουργίας της συγκεκριμένη αρχής. Νομίζω πως ο ρόλος αυτός θα πρέπει να καλυφθεί από κόσμο που έχει απόψεις, ε, όραμα και πεπιθήσεις. Και αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, σας διαβεβαιώ πως ποτέ δεν θα είχα ζητήσει να είμαι υποψήφιος. Θα στη χώρα μου και φυσικά δεν θα τολμούσα να αναλάβω μια τόσο σημαντική θέση. Εγώ πιστεύω πως έχω τις προϋποθέσεις για να ηγηθώ αυτού του προγράμματος. Αναφέρατε επίσης και βέβαια είναι ένας τομέας όπου υπάρχουν αντικείμενα διάφορα συμφέροντα αντικρουόμενα και φυσικά τα εθνικά συμφέροντα. Εγώ αφιέρωσα όλη μου τη σταδιοδρομία στα εθνικά συμφέροντα. 21 χρόνια εργάζομαι στη ρύθμιση και την υποπτία των ασφαλίσεων και των, και ε, ε, συνταξιδοτικών ταμείων. Γνωρίζω λοιπόν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η περάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και είμαι απόλυτα προσιλωμένος αυτό στην εργασία μου. Αναφέρατε τομεί που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή, σε προστασία του καταναλωτή. Είμαι ευτυχή που το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στον κανονισμό αυτό το ρόλο, κατα... την προστασία δηλαδή του καταναλωτή. Νομίζω πω είναι πρόκληση, γιατί όλοι γνωρίζουμε την αρχή τη επικουρικότητα. Είναι πρόκληση, αλλά πιστεύω πω υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και που μπορούν να βελτιωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε έλλειψη ευρωπαϊκής διαδικασίας και στο ε, όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και στις ασφαλείς και στις ε, συνταξιδικά ταμεία. Τι μπορούμε να κάνουμε, συνεργαστούμε με τον κλάδο, με τους ε, διάμεσους, ώστε να εξετάσουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ας πούμε στο θέμα της αποκάλυψης. και νομίζω μάλιστα ότι εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε τα όσα κάναμε στο παρελθόν. Ε, φυσικά ο κόσμος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις ε, σχετικές πληροφορίες, αλλά αυτό που είδαμε στο παρελθόν είναι ότι υπερβολικά πολλές πληροφορίες σκοτώνουν τον καταναλωτή. Θα πρέπει να μιλήσουμε να και να δουλέψουμε για πληροφορίε που είναι σχετικές, που είναι συγκρίσιμες και που αφορούν τα σημαντικά στοιχεία μιας σύμβασης. Τους κινδύνους, ε, τα ασφάλιστρα ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε νομίζω να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές στις χώρες μας για να ε, έχουμε ένα παραπάνω ρόλο στον τομέα αυτό και να βελτιώσουμε την προστασία του καταναλωτή. Τέλος, για τους όρους. Νομίζω ότι φυσικά ο προϋπολογισμός είναι σημαντικός και ελπίζω πως ε, ο προϋπολογισμός θα αυξηθεί ανάλογα με την φιλοδοξία του προγράμματος. Φυσικά θα πρέπει να είναι σταδιακή προσέγγιση, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και επίσης πρέπει να εξετάσουμε και τι ζήτητες που αφορούν τον προπολογισμό. Σίγουρα πολλά μέλη θα έχουν δυσκολία να πληρώσουν το κλειδί 16% για τα επόμενα χρόνια. 60% ε, συγγνώμη για τα επόμενα χρόνια. Αλλά φυσικά και είναι σημαντικό να έχουμε καλό προπολογισμό και καλούς ανθρώπους, γιατί πιστεύω πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που μετράνε ε, και γι' αυτό θα πρέπει να προσλάβουμε ε, τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να συμπληρώσουν αυτούς που ήδη εργάζονται εδώ. Μάλιστα. Και τώρα ο κύριος Κλίντσι. Θα θέλαμε κύριε Μπεραντίνο να έχουμε μια λειτουργούσα ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και, τον, ε, και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξέρουμε ότι όσον αφορά τις ασφαλίσεις και τα συγκεκριτικά ταμεία απέχουμε πόρο από αυτά που θα θέλαμε να επιτύχουμε. Ακόμα πιο άνισος είναι ο τομέας αν δούμε την Αμερική και συγκρίνουμε τη ΣΥΠΑ με την Ένωση. Εσείς βλέπετε να έχει να παίξετε κάποιο ρόλο για να προσπαθήσετε να, ξεπεράσετε αυτές, να ξεπεραστούν αυτές τι διαφορές και να εξασφαλίσετε ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείε θα έχουν κάποια στιγμή πρόσβαση και στις ε, αμερικανικές αγορές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίντς. Είναι μια πραγματικά καλή ερώτηση. δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οριστεί άμεσα. Υπάρχουν ε, πολλά χρόνια πίσω μας με, συζητήσεων με τους Αμερικανούς σε σχέση με, τις, ε, με τους όρους που ισχύουν στις αγορές τους, τις προϋποθέσεις. Αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση. Με το Solvency 2 και με, έχουμε μια δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση στους Αμερικανούς ε, φίλους. Και εγώ δεσμεύομαι βεβαίω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να έχουμε έναν καλό διάλογο με τους Αμερικανούς, ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να υπάρξει βελτίωση όσον αφορά μια σύγκληση, διαδικασία σύγκληση σε όλο το σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πουλήσουμε του Όλμαν τελείω στου Αμερικανού, γιατί δεν πρόκειται να το αγοράσουν σίγουρα. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ένα διάλογο μαζί τους για να εξετάσουμε τους διάφορους τομείς του ρυθμιστικού συστήματος, το κεφάλαιο, τα κεφάλαια, τα διακυβέρνηση και πού μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, για παράδειγμα όσον αφορά την εποπτεία των ομίλων. Είναι αδύνατο να είμαστε ισόμετιμοι με τους Αμερικανούς χωρίς να έχουμε ε, δικό μας εποπτικό σύστημα και θα πρέπει να είμαστε αρκετά δυνατοί εδώ, αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως εγώ θα προσπαθήσω να γυθώ αυτές τις προσπάθειες και να είμαι ξεκάθαρος και όσο δεν δυνατόν περισσότερο διάφανος, εγώ και οι συνάδελφοί μου. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία, γιατί φέρνουμε και τις άλλες χώρες του κόσμου προς την κατεύθυνση μια σύγκληση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Και νομίζω ότι βεβαίως είναι και μια ευκαιρία, όπως σας είπα, να κινήσουμε και τους Αμερικανούς σε αυτή την κατεύθυνση, να περιλάβουμε. Τώρα, ε, στο εκ μέρους του ΕΛΚ, Γκέι Μίτσελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις, συνεχίζοντας ε, το ερώτημα του Βολφ Κλίντς ε, σε σχέση με τη δημιουργία ισότιμων όρων και την προστασία του καταναλωτού. Σε ορισμένε χώρες και στη δική μου έχουμε κοινωνικούς εταίρους που βεβαίως ε, μια σχέση κοινωνικών εταίρων που βεβαίως έχει πολλά πλέον πλεονεκτήματα αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα ε, συνδικάτα ή κυβερνήσεις που τελικά ε, αφήνουν όλοι αυτοί οι αρρώσεις απ' έξω τον καταναλωτή. Πώ προτίθεστε να βάλετε τον καταναλωτή σε μια προεξάρχουσα θέση στην ατζέντα σας. Τώρα, όσον αφορά την επικουρικότητα, μπορείτε να κάνετε κάποιες ε, συγκρίσεις, ε, κάποια στοιχεία σύγκρισης ε, ώστε να, που να μπορείτε να παρουσιάσετε στο Κοινοβούλιο και να υποβάλλετε τις δικές του ερωτήσεις σε σχέση με τη δημιουργία ισότιμων όρων. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της προσθέμενης αξίας και της εφαρμογής, εάν δεν υπάρξει αυτή η προσθέμενη αξία, ποια βήματα θα προτίθεστε να κάνετε και τι κυρώσεις θα επιβάλλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μίτσελ. Βεβαίως οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δική τους φωνή. Και νομίζω ότι η ρύθμιση παρέχει ξεκάθαρες απαντήσεις εδώ, δίνοντας τους ε, καταναλωτές μία ενδεδειγμένη εκπροσώπηση σε όλα τα πάνελ ομιλητών. Νομίζω ότι είμαστε σε μία προνομιακή θέση, γιατί ε, έχουμε το ζήτημα των ασφαλίσεων και των ε, συντάξεων δύο τομείς, ε, δύο πάνελ και θα πρέπει να εκπροσωπούνται και στους δύο οι καταναλωτές για να εκφράζουν τις δικές τους ανησυχίες. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια εκπροσώπηση των καταναλωτών, ούτως ώστε να υπάρχουν ε, πληροφορίες και για μας για τις τάσει τη αγορά ή για τις ανησυχίες των καταναλωτών σε διάφορες χώρες ή για το είδο των προϊόντων που επιθυμούν όπου οι καταναλωτέ επιθυμούν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια οι, οι καταναλωτές θεωρούν ότι ενέχουν ενδυνάμει προβλήματα για το μέλλον. Νομίζω ότι ο ρόλος του πάνελ των ενδιαφερόμενων ε, δεν είναι παθητικός αλλά ενεργητικός. Εξίσου ενεργητικός είναι και ο ρόλος των εκπροσώπων των ε, καταναλωτών. Βεβαίως υπάρχει μια αρχή επικουρικότητας στην οποία άλλωστε αναφέρθηκα, αλλά θα ήθελα να υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική ούτε ώστε η προστασία του καταναλωτού να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα. Και υπάρχουν εδώ πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια ανάλυση για τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την αποκάλυψη κάποιων στοιχείων. Ε, μπορούμε να κάνουμε διάφορες αναλύσεις σε ευρωπαϊκές αγορές προσπαθώντας να εκφράσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και να τα θέσουμε στο τραπέζι. Εγώ βεβαίως θα είμαι και στη διάθεσή σας θα προσέρχομαι εδώ όποτε θέλετε για να ανταλλάσσουμε απόψεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. Τώρα, για το θέμα της εφαρμογής. Αυτός είναι ένας τομέας όπου πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές αποπτικές αρχές πρέπει να ε, δράσουν ε, διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Θα πρέπει να έχουμε τους ιδίους ε, πόρους, ούτως ώστε να ελέγχουμε την εφαρμογή στις διάφορες χώρες μέλη από τις διάφορες εθνικές αρχές. Θα πρέπει να έχουμε τους, ε, ε, δικός μας, ε, τους δικούς μας πόρους. Γιατί ο έλεγχος της εφαρμογής των διαφόρων ρυθμίσεων είναι σημαντικός και θα τον βάλω στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλε Λούντβινγκσον, εκ μέρους του S&D. Σας ευχαριστώ. Ακούω κάποιες ε, ανησυχίες ότι δηλαδή η δημιουργία αυτής της αρχής ε, δεν προχωρά τόσο καλά όσο θα έπρεπε και γι' αυτό και θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την διαδικασία ε, εκκίνησης. Ποιες είναι οι προκλήσεις πιστεύετε όταν θέλετε να οδηγήσετε μια αρχή να δουλέψει σε, με απόδοση 100% ε, και έπειτα έχω κάποιες απορίες όσον αφορά τις πτυχές τις και τους πόρους, τους ανθρώπους που θα χρειαστεί νέα αρχή. Η δική σας άποψη ποια είναι για τους σπόρους που διατίθενται, είναι αρκετή ώστε να μπορέσετε να ασκήσετε το έργο σας σωστά, γιατί εφόσον υπάρχει μια αρχή θα πρέπει να μπορεί και να εκπονεί τα καθήκοντα που τις έχουν ανατεθεί μέσω της εντολής της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λούτβιξον. Ήδη ανέφερα κάποια από τους σημαντικούς τομείς για την εκκίνηση των αρχών. Βεβαίως, τον έχουμε σωστή και στεναρή διακυβέρνηση είναι κλειδί. Κλειδί και για την πολιτιστική, την, την ε, ε, αλλαγή νοοτροπίας που θέλουμε να πετύχουμε. Και νομίζω πως αυτό έχει γίνει τους τελευταίους μήνες και θα συνεχίσει να γίνεται τους πρώτους μήνες ε, του έτους. Για τον προπολογισμό. Εγώ ειλικρινά θα προτιμούσα να είχα ένα ξεχωριστό, μια ανεξάρτητη γραμμή στον προπολογισμό, που να μην τη μοιράζομαι με τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν ήταν αυτή η τελική απόφαση. Φυσικά θα πρέπει να δουλέψουμε με τους πόρους που έχουμε στη διαθεσή μας. Αν με ρωτήσετε αν θα φτάσουν για να κάνουμε όλα τα πράγματα που έχουμε στην αρχή να κάνουμε, θα μου τρελός να σας πω πως ναι. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες, να θεσπίσουμε προτεραιότητες με βάση τους πόρους. Ελπίζω και βασίζομαι στην στήριξή σας ότι θα υπάρξει μια σταδιακή αύξηση του προπολογισμού που θα είναι αντίστοιχη με τη φιλοδοξία του προγράμματος. Είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και πιθανότατα περαιτέρω αλλαγέ και φιλοδοξίες θα προσδεθούν στο μέλλον και φυσικά ο προπολογισμό θα πρέπει να ακολουθήσει, να συμβαδίσει. Εγώ νομίζω λοιπόν πως τώρα θα πρέπει να θεσπίσουμε τις σωστές προτεραιότητες σύμφωνα με τους πόρους που έχουμε και φυσικά να είμαστε δραστήριοι ώστε να υπάρξει μια σταδιακή αύξηση των πόρων μας, πράγμα για το οποίο βασίζουμε στη δική σας βοήθεια. Uh, and... Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα και πάλι εξ ονόματος του ΕΛΚ η Άστρη του Λούλινγκ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε υποψήφι, στην επόμενη ολομέλεια του Στρασβούργου θα ψηφίσουμε για μια ανέκθεση που αφορά το πράσινο βιβλίο της Κομισιόν όσον αφορά την βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών ταμείων. Στις δύο αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπής έχουμε μεγάλες διαφορές απόψεων όσον αφορά ας πούμε το πρόβλημα της ε, την δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων και αν θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί η, οικονομική κατάσταση της κοινωνικής πρόνοιας στον υπολογισμό των κριτηρίων του Μάστρικ, σε σχέση με το ε, δημόσιο έλλειμμα, πράγμα το οποίο συμβαίνει στο Σύμφωνο Σταθερότητας τώρα. Για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο μέσα στο γενικό καθεστώς συντάξεων έχουμε πλεόνασμα. Ένα απόθυμα που επιτρέπει στο κράτος να λέει ότι το έλλειμμα του είναι 1,4% αν λάβει υπόψη όλα τα αποθεματικά. Εάν δεν το ε, παίρνει υπόψη το αυτό θα ήταν στο 3,4% το έλλειμμα. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η δική σας γνώμη και τι θα κάνετε. Και μια τρίτη ερώτηση. Έχουμε και την ε, φερεγγιότητα 2. Άστριντ, συγγνώμη, διακόπτη πρόεδρος. Συγγνώμη. Χρειάζεται και περαιτέρω εγγύησης εκτός από αυτήν την οδηγία στο σύστημα της Solvency 2. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λούλινγκ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Για τις συντάξεις. Ήδη εξέφρασα τη γνώμη μου. Νομίζω ότι με την εξέλιξη του κοινωνικού συστήματος στην Ευρώπη όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένος ρόλος για τον κρατικό ταμείο αλλά και για τα ιδιωτικά ταμεία. Πιστεύω πως είναι δυνατόν να υπάρχει ένα πλαίσιο για την ασφάλεια των συντάξεων στην Ευρώπη που θα μας δώσει περισσότερη προστεθέμενη αξία από ότι μια ελάχιστη, η ελάχιστη εναρμόνιση που έχουμε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να έχουμε, πως πρέπει μάλλον να πάμε στη μάξιμο με εναρμόνιση. Αυτό δεν είναι δυνατόν, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα προς όφελος των εργαζομένων και των καταναλωτών. Αναφέρατε τώρα κάτι άλλο, την δυνατότητα μεταφοράς. Ναι, φυσικά αυτό θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο οποιοδήποτε συνταξιδοτικού συστήματος. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως πρόκειται και πολιτικό ζήτημα στην Ευρώπη. Στο παρελθόν έγιναν απόπειρε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό, είναι πολιτική απόφαση. Εγώ νομίζω πως είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε ένα συνταξιδοτικό σύστημα. Και αν κανείς εξετάσει το σύνολο της οικονομίας στην ανάγκη, ανάπτυξη στην ανάγκη, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, νομίζω πως θα παίξει αυτό σημαντικό ρόλο. Bring to the table uh, on the pensions area, it's um, the, future of pensions. Τώρα, το μέλλον των συντάξεων καλεί να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε δύο πράγματα. Δηλαδή, από τη μια πλευρά ε, σύνταξη για όλους, αλλά και προσιτές τιμές. Η πρόκληση είναι αυτή. Να συνδυάσουμε και τα δύο. Δεν μπορεί να υπάρχουν free, ε, ε freelance. Η προστασία έχει μια τιμή. πρέπει απλώ να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Και εδώ νομίζω πως υπάρχει και χώρος για καλύτερη μοιρασιά των κινδύνων ανάμεσα στα μέλη, τους δικαιούχους, αλλά και τις χρηματοπιστωτικές αγορές που πρέπει να βελτιωθούν και να δώσουν καλύτερες λύσεις στην ασφάλεια για τη συντάξη στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε χρόνο και για μία ακόμη ερώτηση. Φιλελεύθερη, τρεμόσα, οραμών. θα χρησιμοποιήσω το εναπομένον λεπτό για το επόμενο θέμα, για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Αλλά ο Πασχάλης να μιλήσει τώρα. Μάλιστα, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Χαίρετε. Εγώ το εναπομένον λεπτό θα το χρησιμοποιήσω για να θέσω το ερώτημα που είχα θέσει και στον προηγούμενο δηλαδή στον υπεύθυνο της ΕΑΚΑ, ε, το σύνολο των πρακτικών των συναντήσεών σας με εκπροσώπους της βιομηχανίας το έχετε δημοσιεύσει όπως έγινε ζητήθηκε από τις Ηνωμένε Πολιτείες ώστε οι κοινοβουλευτικοί και οι κοινοβουλευτικές να μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς είπατε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Πρέπει να σεβόμαστε τους κανονισμούς και ό,τι αυτοί προβλέπουν. Προβλέπει δε αυτός ο κανονισμός ότι όλες οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των ενδιαφερομένων θα δημοσιεύονται. Και φυσικά θα δημοσιεύονται και θα γίνονται, θα διατίθενται. Κατά τη δουλειά μου θα κάνουμε φυσικά επίσημες και ανεπίσημες συζητήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες γιατί εγώ πιστεύω στην απόλυτη διαφάνεια. Γιατί νομίζω ότι προσθέτει πολλά είναι πολύ ωφέλιμη. Αφού λοιπόν το προβλέπει ο κανονισμός, δεν είναι για μένα πρόβλημα να δημοσιεύονται οι συζητήσεις αυτές και να σας έρχονται δεόντως. Να ακουστούν και να τυπωθούν όλα. Δεν το θεωρώ προβληματικό. Βέβαια, οι απόψεις των εκπροσώπων της βιομηχανίας χρειάζονται ειδική άδεια για να δημοσιευτούν. Ειδική εντολή. Γιατί, διότι αν υπάρχουν άτυπες συνεννοήσεις μεταξύ της αρχής και της βιομηχανίας, οι κανόνες καλής συμπεριφοράς θα πετούσαν να δημοσιευθούν αυτά εφόσον συμφωνούν όλοι. Εγώ είμαι υπέρ της δημοσίευσης και της διαφάνειας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μυστικότητα σε τέτοιες συζητήσεις. Γι' αυτό, αν το λέει ο κανονισμός, εγώ θα ήμουν υπέρ, υπέρ της δημοσίευσης των πάντων. Δεν, εφόσον δεν πρόκειται βέβαια για εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συζητήσει η ανταλλαγή απόψεων δεν έχουν πρόβλημα. Μάλιστα, σας κατευχαριστούμε. Τελειώνει και αυτή η ακρόαση. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Μπορείτε να αποχωρήσετε. Ο Γαβριήλ εννοώ, οι άλλοι να μείνουν και οι άλλες γιατί θα γίνει και η τρίτη και τελευταία ακρόαση. Δύο λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παρακαλώ, είπα υπάρχουν θέσεις πίσω. Προχωρείτε στο διάδρομο να ξαναρχίσουμε. Μάλιστα. Τώρα κάνουμε την τρίτη και τελική μας ακρόαση με τον Ανδρέα Ένρια επιλεγέντα υποψήφια τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ΕΑΤ. Σας ξαναυπενθυμίζω τη διαδικασία γιατί ορισμένοι προσήλθαν τώρα. Πρώτον ο κύριος Ένρια θα μας κάνει μια παρουσίαση πεντάλεπτη, μετά θα αρχίσουν οι ερωτήσεις απαντήσεις Ένα λεπτό για την ερώτηση, όχι πολύπλοκες ούτε πολλαπλές ερωτήσεις γιατί αυτό είναι άδικο και οι απαντήσεις σε 3,5 περίπου λεπτά, το πολύ σύνολο 5 λεπτά ερώτηση και απάντηση. Μέχρι τώρα πήγε πολύ καλά το σύστημα αυτό. Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή λοιπόν δίνω το λόγο στον Ανδρέα, στον κύριο Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Η ίδρυση αυτής της καινούργιας αρχής σημαίνει, σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή. Χρειάζεται μια αλλαγή, περισσότερη εποπτεία. Είναι δύσκολο βέβαια να επιτευχθεί σύγκληση στην εποπτεία αλλά την άνοιξη του 7, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει η κρίση, θυμάμαι ότι είχαμε δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μιας μελέτης για την επιτευχθήσα μέχρι τότε πρόοδο στην εποψία και ήταν και μερικοί από εσά που είχαν πάρει μέρος και αυτό ήταν πολύ σημαντική στιγμή. Οι περισσότεροι που συμμετέσχουν στη μελέτη εκείνη επένεσαν τη δουλειά της ΣΕΜΣ διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους, διαβουλεύσεις, αλλά επίσης οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν παρατήρησαν καμία επίπτωση στην καθημερινή πρακτική των εποπτικών αρχών. Με το ξέσπασμα της κρίσης φάνηκε ακόμη περισσότερο πόσο αρνητικό ήταν αυτό. Γιατί εθνικά κυρίως ζητήθηκε απάντηση στην κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε καινοτομίες για να αλλάξει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα έχει περισσότερες δικαιοδοσίες από την προηγούμενη εποπτική αρχή. Γνωρίζω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόκληση. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Αυτό που μπορώ να σας προσφέρω εγώ εάν εγκριθώ ως πρόεδρος είναι να οικοδομήσω, να προσπαθήσω να οικοδομήσω μια πραγματικά ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Από την καριέρα μου στο ΣΕΜΣ και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπόρεσα να συμβάλλω στην λήψη ορισμένων αποφάσεων που βλέπω ότι είναι πολύ χρήσιμες. στην Κεντρική Τράπεζα, το Μάζο Παλασκιώπα, τον είχε κάνει για πρώτη φορά την πρόταση για ενιαίους κανόνες εποπτείας. Ξέρω ότι δεν θα πετύχει αυτό το νέο πλαίσιο παρά μόνον εάν υπάρχουν πραγματικές δικαιοδοσίες της αρχής αυτής. μάλλον θα σημειωθούν περισσότερες διαμάχες. Γιατί δεν επιζητούμε πάση θυσία συνένεση. Επιζητούμε ποιοτική δουλειά. Το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει τα εργαλεία. Οι οικειοδοσίες της ΕΑΤ είναι ευρείες. Πρέπει να καθορίσει προτεραιότητες και να διαχειριστεί τις προστοκίες όλων των ενδιαφερομένων πρώτη από τις οποίες πρέπει να είναι η επιτυχία του, των ευρωπαϊκών δοκιμών ε, κρίσεων ή στρες. ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα εάν χρειαστεί. Δεύτερον, η ΕΑΤ πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί όντως να κινηθεί με ενιαίους κανόνες. Εξάλλου και τον περασμένο Νοέμβριο στη Σεούλ το ΓΑΜΑ 20 περίπου αυτά είπε. Πρόκειται για θέματα που δεν πρέπει να, να χαρακτηριστούν από ρυθμιστικό ανταγωνισμό. Δεν αρκεί λοιπόν να παραμείνουν κατακερματισμένες, κατακαιρματισμένα τα προγράμματα εποπτείας χωρίς να γίνει ένας πραγματικός συντονισμός τους. Και πρέπει οι κανόνες της ΕΑΤ να γίνουν κατανοητοί από τους τελικούς χρήστες και χρήστριες, ώστε να υπάρξει και προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών, όπως προβλέπει η Κομισιόν για την ενιαία αγορά. Τέλος, η ανεξαρτησία των αρχών αυτών είναι σημαντική και από τη βιομηχανία για να μην υπάρξει επηρεασμός και από τα άλλα θεσμικά όργανα για να μην στρεβλωθεί η πολιτική της και έτσι η θέση σε κίνδυνο του χρηματοπιστωτικού σύστημα. Επίσης όμως χρειάζεται να είναι και υπόλογη αρχή. Εάν εγκριθώ θα συνεχίσω το διάλογο με την Επιτροπή σας, την Πρόεδρό σας και τα μέλη σας. Επίσης νομίζω πρέπει τακτικότερα να γίνονται συνεννοήσεις και ανταλλαγές απόψεων με τους βουλευτάς. Ευχαριστώ πολύ και θα ακούσω με τα χαρά στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Η πρώτη εκ μέρους του ΕΛΚΑ από τον Μπέρκχαρτ Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ενερία, βρίσκω ότι έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία και αυτή τη στιγμή είστε επικεφαλής της, ε, ε, της στη Ρώμη. Ε, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε και προς τους άλλους ε, υποψηφίους. Αναφερθήκατε ήδη σε αυτό. Πώς θέλετε να εξασφαλίσετε πραγματικά την ανεξαρτησία της αρχής σας και ποια είναι η δυνατότητα επιβολής δική σας έναντι των εθνικών εποπτών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να διατηρούν τα δικά τους δικαιώματα. Τέλος, είπατε ότι θέλετε να έχετε έναν ενεργητικό διάλογο μαζί μας. Πώς το φαντάζεστε, μπορείτε να μας ε, πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Yes, thank you. Ναι, σας ευχαριστώ. Η ανεξαρτησία είναι το κλειδί, όπως είπα. Η ανεξαρτησία από τις εθνικές αρχές βεβαίως είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, γιατί ε, το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα, πρέπει να συμμετέχουν οι εθνικές αρχές. Αυτό το οποίο έλεγα στην ε, συνέντευξη με το Συμβούλιο ε, Εποπτών, εδώ υπάρχει μία σημαντική διαφορά γιατί αν δείτε το ρόλο των εθνικών εποπτών βλέπετε ότι συζητήσαν να τα ονόματά τους αλλά και η χώρα προέλευσης. Δηλαδή παρόλο που επιλέγονται οι άνθρωποι αυτοί ε, τώρα ως προερχόμενοι από τις χώρες μέλη αυτή τη στιγμή θα είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο θα εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια συμβολική αλλαγή. Ε, η οποία θα αντανακλάται και στην ιδιότητά τους πλέον, στην νέα τους ιδιότητα. Ε, μέχρι τώρα υπήρχαν επιτροπές εμπειρογνωμόνων, δηλαδή οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες προετοίμαζαν το τεχνικό έργο και συνήθως αυτή είναι, ε, αφήσατε περισσότερο στις αλλαγές οι μας σε εθνικό επίπεδο, γιατί είναι συνηθισμένοι να κάνουν τα πράγματα όπως τα έκαναν πάντα. Συνεπώς λοιπόν, όταν έρχονται στο τραπέζι ιδιαίτερως ε, ευαίσθητα πολιτικά θέματα, είναι σημαντικό ε, οι άνθρωποι αυτοί να εξασφαλίσουν κάποιες, ε, να, να είναι σημαντικό να εξασφαλίσουν κάποιες αλλαγές και σε, που να φτάνουν και στο εθνικό επίπεδο, στο επίπεδο των εθνικών εποπτών. Στην ε, Ιταλία, στην, ε, εγώ δούλεψα στην Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, η οποία δίνει, όπως ξέρετε, μεγάλη σημασία στην αυτονομία της, στην ανεξαρτησία της. Και ε, θεωρώ και εγώ ότι η ανεξαρτησία στην κρίση και στην αξιολόγηση του τι συνιστά ακριβώς την δημόσια ωφέλεια την οποία εξυπηρετούμε, το δημόσιο συμφέρον βρέθηκα και στο παρελθόν σε καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που υπήρχαν συγκρούσεις συμφερόντων συγκρούσεις συμφερόντων με την Τράπεζα της Ιταλίας όταν εγώ ήμουνα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ποτέ η Τράπεζα της Ιταλίας δεν με πίεσε για να εκπροσωπήσω μια εθνική προοπτική ή τις, ε, να προσπαθήσω στις εθνικές θέσεις και ποτέ δεν το έπραξα όταν ε, ήμουν πεπισμένος ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ήταν διαφορετικά. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βεβαίω υπάρχουν ήδη πάρα πολλά εργαλεία στη δική σα ε, νομοθεσία που ήδη υπάρχουν και μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα όποτε θέλετε και ασφαλώ θα έρθω και θα μαζί σα. Αλλά θα ήθελα να σα πω ότι το έργο της ΕΑΤ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, θα είναι εξαιρετικά διαφανές. Δηλαδή, όποτε προετοιμάζονται κάποια σχέδια κανονισμών, θα ε, προηγηθούν δημόσιες ακροάσεις, θα δημοσιευθούν τα κείμενα στο website κλπ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ερώτημα εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, εκ μέρους του κυρίου Σάντσεθ Ποσέδο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω να σας καλωσορίσω σε αυτή την Επιτροπή. Για πρώτη φορά έχουμε μία, έναν υποψήφιο εδώ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Συνήθως είναι μια σημαντική στιγμή. Είπατε σε σχέση με το ρόλο του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ε, δεν θέλουμε απλώς ε, να λαμβάνετε υπόψη σας την ε, γνώμη μας. Είναι πολύ σημαντικό να μας εγγυηθείτε μια αποτελεσματική ηγεσία ούτως ώστε να καταστεί εφικτό το αναγκαίο. Ε, ε, ε, σε λίγο καιρό θα πρέπει να ανταποκριθείτε στα τεστ αντοχής. Ξέρετε, τα προηγούμενα τεστ αντοχής εμφάνισαν κάποια προβλήματα. Θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα σε σχέση με το τι ακριβώς απέτυχε και τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η αποτυχία στο μέλλον. Πραγματικά το βιογραφικό σας είναι ιδιαίτερος ε, ικανοποιητικό όσον αφορά τον ευρωπαϊκό συντονισμό και μια προ... Ε, κυκλική ε, πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρεσέδο για αυτή την ερώτηση. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. χρειάζεται να επιδείξω μια στεναρή ηγεσία ένα ηγετικό προφίλ ε, στον τομέα αυτό. Ε, είναι σημαντικό να αποδείξω τη δέσμευσή μου υπέρ του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Εγώ έχω δουλέψει στο παρελθόν σε επιτροπές περιβάλλοντος και ε, το θέμα είναι ότι σημαντικό είναι όταν πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση ορισμένων διαφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιδιότητα, η ικανότητα διθέτηση των ε, διαφορών. Ε, και νομίζω ότι εγώ την έχω αποκτήσει από την εμπειρία μου. Έχετε δίκιο όταν ε, λέγεται ότι το πρώτο τεστ επιτυχίας θα είναι το τεστ αντοχής των τραπεζών, για να κάνω αυτό το λογοπαίγνιο. Το stress test, το τεστ αντοχής θα είναι είναι στο στο θέμα. Νομίζω και επιτρέψατε μου να πω ότι τα τεστ αντοχής δεν, είναι, δεν έχουν την αξία της πρόβλεψης. Ναι, μεν ε, καταλήγει κανείς σε κάποιο αποτέλεσμα και στη συνέχεια ε, μπορεί να πει ότι οι εξελίξεις στην αγορά τους επόμενους ε, μήνες τελικά είναι δυνατό να θέσουν να τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής, της δοκιμής αντοχής για παράδειγμα αυτό το οποίο έγινε το περασμένο καλοκαίρι από τη ΣΕΠΣ, όπου είχε ε, ε εκπονηθεί ένα σοβαρό σενάριο το οποίο είχε λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, ένα αρκετά σκληρό σενάριο αλλά στην πραγματικότητα δεν υλοποιήθηκε στη συνέχεια και μπορούν να υπάρχουν εξελίξεις σε ορισμένες χώρες πολύ πιο ε, σκληρές από αυτό το οποίο έχει προβλέψει το τεστ αντοχής. Για παράδειγμα αυτό το οποίο έγινε στην Ιρλανδία. Και βεβαίως αυτό έδωσε ε, λαβή σε διάφορα θέματα χρηματοδότησης, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη διάφορα τεστ αντοχής αλλά αξιολογούν περισσότερο τους πιστοτικούς κινδύνους. Ε, νομίζω ότι αυτό το χρόνο θα πρέπει να έχουμε μια πιο... Ε, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία και ισχύ. Νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις τομείς όπου θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτον, μεθοδολογικά ότι πέρσι ε, είχαμε την εντολή μιας εσωτερικής εποπτικής λειτουργίας η οποία δεν ε, πρόκειται να κοινοποιηθεί. Φέτος θα κοινοποιηθεί η εποπτική μας ε, λειτουργία, θα διατυπώσουμε τις προσδοκίες μας στους διάφορους οίκους αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, στους συμμετέχοντες κλπ. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί από ότι το περασμένο έτος. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των τραπεζών. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστα εργαλεία που να διασφαλίζουν αυτή την συνοχή, τη συνέπεια μεταξύ των διαφόρων τραπεζών γιατί πέρσι είχαμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ τραπεζών με παραπλήσια χαρτοφυλάκια. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτή τη ε, συνοχή, τη συνέπεια. Ο τέταρτος ε, τομέας αφορά τη ρευστότητα, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ε, δεν ήταν να εξασφαλίσουμε, να προβλέψουμε ρευστότητα και αξιολόγηση του κινδύνου εντός του ιδίου τεστ αντοχής θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε και το, την πτυχή της ε, ρευστότητας εξίσου. Σας ευχαριστώ. Επόμενος, εξ της ομάδας Άλντε, η, Σιλβί Καλημέρα σας. Μιλώσατε, μιλήσατε για τον Τομάζο Παντοσκιώπα και φαντάζομαι πως ε, θα είστε πιο θλιμμένος από ότι εγώ για, που δεν βρίσκεστε στο Μιλάνο στο Πανεπιστήμιο Μποκόνη για να τιμήσετε τη μνήμη του. Πάντως νομίζω πως και εμείς με τον τρόπο μας τιμούμε την μνήμη του. Μιλούσε για τα καρτέλ των εθνικισμών εκείνος. Ήταν μια αγαπημένη του ρίση. Εσείς τι θα κάνετε και αυτό αφορά εσά αν και έθεσα και την ερώτηση αυτή στον κύριο Μαγιόρ ε, πριν από λίγο και τα είδαμε τα κράτη-μέλη, δεν πρέπει να αυτοπατώμεθα, δεν ήθελαν, τουλάχιστον όχι όλοι, πολύ ευρωπαϊκή και ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποπτήρια, γιατί αυτό θα του ενοχλήσει στο, οι σχέσει του με τον τραπεζικό τομέα για τα πράγματα που δεν πάνε καλά. Όταν θα προσπαθήσουν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν το άρθρο 23 που εφήβραν για να βάλουν ένα, μια σούπερ κλειδαριά στην δική σας ε, εξουσία και όταν θα λάβουν αποφάσεις που θα έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις βαριές για κάποια κατημέλη, εσείς τι θα κάνετε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ερώτημά σας, ε, την ερώτησή σας και για την αναφορά που ε, που κάνατε στη δουλειά του Τομάζο Παλουσκιάπα. Όντω θα αποτελέσουν οι εργασίε του έναν οδηγό για μας. Καταρχήν μετακινούμαθε από έναν κόσμο συνένεσης και ομοφωνίας προς ε, μία ε, δομή που θα υπάρχουν ψηφοφορίες και μάλιστα θα πρέπει κανείς να αναλάβει προσωπικά ευθύνη σε κάποιες ε, περιπτώσεις. Αυτό ήδη βοηθά στο να φτιαχτεί μια πιο ε, ευρωπαϊκή μορφή και σώμα και ότι, ώστε ο κόσμος να αισθάνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να δράσει κανείς σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεύτερον, νομίζω ότι υπάρχει μια άλλη μεγάλη διαφορά, ότι αυτή τη στιγμή αποδίδονται εξουσίες στην αρχή που δεν υπήρχαν παλιότερα. Άρα πρέπει να είναι σαφές πως ε, αυτές οι αρμοδιότητες θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν τρεις τομείς και χάρη στην εργασία του Κοινοβουλίου όπου οι αρχές ε, έχουν δυνατότητες να ξεπεράσουν τις αποφάσεις των εθνικών αρχών. Πιστεύω πως ε, δεν θα υπάρξει λόγος να τα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα ή εν πάση περιπτώσει όχι συχνά, αλλά το γεγονός ότι τέτοιες, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες δίνει αυτό μεγαλύτερη ισχύ στην ευρωπαϊκή προοπτική ώστε να αποφύγουμε τα εθνικά συμφέροντα να μπλοκάρουν και να εποδίσουν την πρόοδο. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα οι εθνικές αρχές να εκφράσω ανησυχίες. Φαντάζομαι πως αναφερόσαστε στην δημοσιονομική ρήτρα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η αρχή να ενεργήσει σαν να μην υπήρχε αυτή η ρήτρα. Να αποφασίσουμε δηλαδή ποιο είναι το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και έπειτα όντω μπορεί να υπάρξουν περιπτώσει όπου μπορεί ένα κράτο μέλο να θεωρεί πω παρεμβαίνουμε στην εθνική κυριαρχία και είναι καλό να υπάρχει ένα εργαλείο στο θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θίγουν αυτό το θέμα και να το φέρνουν προς συζήτηση. Και να υπάρχει και διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων, γιατί έτσι τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα και δεν ασχείται πίεση ώστε να απομακρυνθούμε από τις αρχικές αποφάσεις. Αυτό που ήταν σημαντικό και το Κοινοβούλιο μέσα στον κανονισμό έκανε καλή δουλειά και το εμπόδισε αυτό, είναι να μην φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ως εποπτική αρχή, αν πάμε δηλαδή προς τα πίσω, να υπάρχει πάντοτε ένας δημοσιονομικός αντίκτυπος, γιατί είμαστε εκεί για να ε, ε, ε, αποφύγουμε τις κρίσεις και τον αντίκτυπο των κρίσεων στους φορολογούμενους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος αιτιολογημένος πίσω από τα εθνικέ εθνικές ανησυχίες και όχι μόνο το ότι μπορεί να παρεμβαίνει στην εθνική παρε... Ε, εποπτεία, γιατί αυτό θα κάνουν οι αρχή αυτή. Ευχαριστώ. Και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων ο Σβέν Κίγκολτ. Μάλιστα. Χαίρετε. Καταρχήν χαιρετίζω το στεναρό ευρωπαϊκό πνεύμα που εκφράσατε. Είναι ευχάριστη διαφορά με ορισμένους προηγούμενους. Δεύτερον, με ενδιαφέρει πολύ να δω πώς θα χρησιμοποιήσετε τη δικαιοσία σε δύο τομείς. Ένα, πώς θα διασφαλίσετε ότι τα εκτός ισοζυγίου τμήματα της τραπεζικής δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη. Ξέρετε ότι πολλές φορές έχει γίνει λόγος για σκιώδεις τράπεζες. Πώς θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν τις δικαιοδοσίες σας ώστε να αποσαφινιστεί ότι θα υπάρχουν όλα στην εποπτεία. Και δεύτερον, για την προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών, πώς θα διασφαλίσετε ότι οι τράπεζες θα εργάζονται καλύτερα όταν ε, εξυπηρετούν μικροπελάτας. Ευχαριστώ. Τα ερωτήματα αυτά είναι πολύ λεπτά. Για τα θέματα off balance sheet, εκτός του, του επισήμου ισοζυγίου της τράπεζας. θα προσπαθήσω να υπάρξει συνεπής και ομοιόμορφη συμπεριφορά των προϊόντων και διαδικασιών εποπτείας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες έκαναν τα ισολογισμούς τους. Τους Αλλά και αυτό δεν αφορά καθαρά την εποπτεία, είναι το λογιστικό μέρος. Εγώ θεωρώ ότι οι περισσότερες από τις σκιώδεις λεγόμενες δραστηριότητες θα έπρεπε να είχαν τεθεί υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών. Υπάρχει λοιπόν κάτι που μπορεί να κάνει το ενιαίο εποπτικό πλαίσιο. Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα είναι πρόβλημα Ξέρουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα αυστηρότερα για τις τράπεζες, γιατί αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα του γάμα 20 της Σεούλ. Αυξάνοντας λοιπόν τις απαιτήσει μας από τις τράπεζες, μειώνουμε τους κινδύνους και για άλλα τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρέπει άρα να υπάρξει μία συνεπής και συνολική προσέγγιση για όλα αυτά. Η ESRB θα το προσέξει αυτό. Προσέξει. Και εγώ αν είμαι ο πρόεδρος στη ΣΕΑΤ θα το προσπαθήσω. Ξέρουμε ότι όποτε σημειώνεται κάποιος κίνδυνος, τότε σε περίπτωση κρίσης χρειάζεται τελικά να δοθούν ρευστά για να βοηθήσουν τις τράπεζες. Άρα η συμπερίληψη όλων των δραστηριοτήτων στον ισολογισμό είναι κάτι το ζωτικό ώστε να γνωρίζουμε ποιες δραστηριότητες μπορεί να καταλήξουν στη δημιουργία κινδύνου ή κρίσης. Όσο για τη προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών, στο παρελθόν δεν ξέρω αν υπήρξε καμία τέτοια επιτυχία, αν μπορούμε να πούμε. Έχουμε ένα προσωρινό πρόγραμμα λειτουργίας της ΕΑΤ που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα στοιχείο προστασίας καταναλωτριών. Αλλά επειδή είναι προσωρινό δεν θα έπρεπε να το σχολιάσω τώρα, δεν θα ήταν πρέπον. Προσωπικά όμως, προσωπικά, νομίζω ότι υπάρχουν τομείς όπου ήδη η Κομισιόν ασχολείται με θέμα προστασίας καταναλωτών και καταναλωτριών, responsible landing και άλλα, και από ό,τι βλέπω από την εθνική εμπειρία των κρατών από έγγραφα της Κομισιόν στην ιστοσελίδα της υπάρχουν τουλάχιστον δύο τομείς όπου θα ήθελα να γίνει ακόμη πρόεδρος. Ο ένας είναι η διαφάνεια για τις συνθήκες που εφαρμόζονται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για τις καταθέσεις γιατί στην Ιταλία τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει προστασία του καταναλωτή γι' αυτό. Και δεύτερον, ο καθορισμός περαιτέρω διευκολύνσεων για τη διαφορα... επίλυση διαφορών μεταξύ πελατών και τραπεζών. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω, όχι άσχετες ερωτήσεις πάνω από μία δηλαδή. Ο Πασχάλης δεν θα ξαναμιλήσει. Ευχαριστώ που μιλήσατε, που κάνατε λόγο για την δοκιμή αντοχής του καλοκαιριού. Έγινε επιτυχώς η δοκιμή και μετά λίγους μήνες μετά οι, τραπε... Ιρλανδικές τράπεζες κήρυξαν σχεδόν πιτόχευση. Δεν ξέρω λοιπόν ποιο είναι, ποια είναι η ποιότητα των δοκιμών αυτών και ζητήθηκαν και άλλες εξαιρέσεις και από ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες. Ίσως ορισμένοι να προσπαθούσαν να προστατεύσουν ορισμένες τράπεζες ακόμη και κατά τη διενέργεια της δοκιμής. Πώς θα αποφευθεί κάτι τέτοιο αν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να αποκλείονται οι δικές τους τράπεζες από τα μέτρα προστασίας και ιδιαίτερα οι εξαιρέσεις που χορηγούνται στα ψηλά των οδηγιών θα ισχύσουν. Εσείς θα είστε και υπέρ των τραπεζών και υπέρ των πολιτικών. Πώς θα τα συνδυάσετε. Ευχαριστώ για την δοκιμή αντοχή σας. Είχα υπονοήσει ήδη προηγουμένως ότι ότι Πράγματι ήταν απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Ποιοι είναι οι λόγοι όμως. Θέλω να τους πω. Πρώτον, τα κριτήρια της δοκιμής ήταν το 6% τον πρώτο χρόνο, ενώ τα κεφάλαια που απαιτούνται τώρα για τις Ιρλανδικές τράπεζες λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων που ισχύουν εκεί είναι πολύ ψηλό το διπλάσιο 12% τα κριτήρια αυτά είναι λοιπόν και υπήρξε και ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόβλημα των Ιρλανδικών τραπεζών όποτε το ρευστό μιας τραπέζης λείπει, τότε λείπει και η αξιοπιστία προς αυτήν. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να είναι πιο αυστηρή η δοκιμή αντοχής και να υπάρξουν και επαληθεύσεις μεταξύ εποπτών για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Όχι μόνο το περιεχόμενο των εθνικών δοκιμών αντοχής. Για τις εξαιρέσεις τώρα Πιστεύω ότι χρειάζεται να ληφθούν υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών τραπεζικών αγορών. Στους κανόνες της Βασιλείας ας πούμε. Νομίζω ότι οι εθνικοί επόπτες ήδη είχαν καταφέρει να συζητηθούν στη Βασιλεία ορισμένες ιδιαιτερότητες όπως τα, κεφαλ... τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες ή δίκτυα. Αυτά ήδη τα λέει το κείμενο της Βασιλείας, αλλά πρέπει και να εφαρμοστούν με τις λεπτομέρειες τους στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως προς την ειδική έτερη αναγνώριση εξαιρέσεων ειδικών μεταχειρήσεων κλπ. στο παρελθόν και εγώ και οι ΣΕΜΣ ήμασταν πάντοτε κατά των εξαιρέσεων και πρέπει αυτή τη φορά να το πετύχουμε. Όσο περισσότερο εσείς και το Συμβούλιο θα συμφωνείτε επί των προτύπων χωρίς εξαιρέσεις, τόσο το λιγότερο θα υπάρχει το πρόβλημα αυτό διαφορετικής μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων εξ ονόματος του ΕΛΚΟ, Ότμαν Κάρας. Ναι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις μέχρι τώρα. μιλήστε για τις αρμοδιότητες σας και ταυτόχρονα για τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις προκλήσεις και το Single Rule Book. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Έχετε αρκετές αρμοδιότητες για να υλοποιήσετε αυτό το οποίο εξαγγείλατε ότι προτίθεστε να κάνετε. Πού χρειάζεστε μια πλήρη εναρμόνιση σε σχέση με το Single Rule Book. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Πού βλέπετε ότι αποσιάζουν συνολικές ε, ρυθμίσεις για να μπορέσουν να δημορφώσουν αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή εποπτεία σε ένα παγκόσμιο ε, πλαίσιο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καράσα και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω επίσης και για όλη την εργασία που κάνατε ε, στο σχέδιο έκθεση για το CRD4, το οποίο εκτιμώ πολύ. Το ερώτημά σας κατά πόσο έχω πράγματι τις εξουσίες τις οποίες χρειάζομαι για να τα εφαρμόσω όλα αυτά. Νομίζω ότι ότι στο κανονισμό προβλέπονται ισχυρές αρμοδιότητες και αν είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, το καθήκον μου θα είναι να αξιοποιήσω αυτές τις εξουσίες, να χρησιμοποιήσω αυτές τις εξουσίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ούτως ώστε να εξασφαλίσω μια πρόοδο. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ενδειγμένο τώρα να πω ότι θα έπρεπε να έχω περισσότερες εξουσίες ότι δεν έχω αρκετέ εξουσίε για να ε, πετύχω, να σημειώσω κάποια πρόοδο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τη ρύθμιση αυτή, ε, να λειτουργήσει δυνατόν καλύτερα και να εξαντλήσουμε το δυναμικό το οποίο προσφέρει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Όσον αφορά το single rule book στο οποίο αναφερθήκατε, τόσο στην ε, ρύθμιση όσο και στο έργο που έχει γίνει στην οδηγία Omnibus, ε, νομίζω ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τομέων όπου θα υπάρξουν κοινοί κανόνες και θα ήθελα να ξεπίσω την ευκαιρία αυτή για να πω κάτι σε σχέση με το Single Rule Book. Ε, πίστευα πάντοτε ότι δεν αφορά μόνο το, ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ενιαίο κανόνα ε, που να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά επίσης και την ε, ορατότητα, το βαθμό ορατότητας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε, σύγκριση με την, σε σχέση με την εθνική νομοθεσία. Μέχρι τώρα έχουμε φτιάξει πολλές οδηγίες που είναι σημαντικές, αλλά όσον αφορά τις τράπεζες, όταν πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες, αυτό το οποίο είναι σημαντικό για αυτές είναι η εθνική νομοθεσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ορατότητα για το πραγματικά ευρωπαϊκό τμήμα της νομοθεσίας. Ε, νομοθεσίας. Ορισμένες φορές όπως λέω, ασκώντας το επάγγελμά μου, διαπιστώνω πολλές φορές ότι οι εθνικοί ρυθμιστές κατηγορούν τις ε, Βρυξέλλες διότι βάλουν εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες ε, στον τομέα αυτό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι τράπεζες ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες και επιπλέον θα υπάρξουν κάποιοι άλλοι κανόνες που απαιτούνται σε ορισμένους τομείς για να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες δημορφίες των εθνικών αγορών. Και βεβαίως τα όρια μεταξύ των δύο θα πρέπει να είναι κινητά. Το βεβαίως ο ευρωπαϊκός γνώμονας είναι καθοριστικός και το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα είναι ευρύτερο ε, από αυτό που είναι σήμερα. Ανέφερα στα εισαγωγικά μου λόγια το θέμα της ρευστότητα, την ε, υποχρέωση αναφοράς των εποπτικών αρχών ε, και διαφορά άλλα. Ε, υπάρχουν κάποιες δεσμευτικές προδιαγραφές στην διαδικασία αυτή που νομίζω ότι συνεπάγονται μεγάλο φόρτο εργασίας για μας. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών τώρα, ο Τζιάννη Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ενερία, εσείς ως, ως επικεφαλής της ρύθμισης της Τράπεζας της Ιταλίας, καθώς και λόγω της αξιοπιστίας που έδειξε το χρηματοπιστωτικό ιταλικό σύστημα κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης, αποτελέσατε ένα από τους, έναν από τους ανθρώπους κλειδί στο πλαίσιο της Επιτροπής για τη Βασιλεία που καθόρισαν το νέο πλαίσιο πρόληψης που καθορίζεται από την Βασιλεία 2 και θα οδηγήσει η Βασιλεία 3. Δραματικές ε, επιπτώσεις κινδυνεύει να έχει η Βασιλεία 3 στο επίπεδο της χρηματοδότησης της οικονομίας που θα περιοριστεί κυρίως λόγω και μάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορείτε να μας δώσετε την αποψή σας σε αυτό το θέμα και τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει η ΕΜΠΑ όσον αφορά την ε, αποκλιμάκωση των αρνητικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πιτέλα. Αν δεν σας πειράζει θα απαντήσω στα αγγλικά. Ξέρω πως υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις επιπτώσεις της Συμφωνίας Βασιλεία 3 και τη χρηματοδότηση της οικονομίας και των ΜΜΕ, μικρομεσαίων δηλαδή, ε, όλος ιδιαίτερος. Η έκθεση του κυρίου Κάρας, το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κάρας για την ε, CRT4 ήδη περιλαμβάνει αυτές τις ανησυχίες και τις εκφράζει να σας πω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά για να μετρηθεί και να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων στις τράπεζες και στην χρηματοδότηση της οικονομίας. Η ΣΕΠΣΕ το Δεκέμβριο δημοσίευσε μια μελέτη, συνολική μελέτη για 246 τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το αποτέλεσμα είναι πως αν δει κανεί το σύνολο των απαιτήσεων, δηλαδή 4,5% μίνιμουμ απέτηση για τις, τα κοινά χρεόγραφα, συν ε, το 5% της συντήρησης κεφαλαίων, του συγκεκριμένου φράγματος κεφαλαίου, ναι. οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα είχαν στο τέλος του 2009 ένα έλλειμμα 209 δις. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό που, ε, ανησυχούν, που ανησυχείτε μάλλον για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Θα πρέπει να σας πω ότι η αντίκτυπος ήταν βασικά για τις μεγαλύτερες τράπεζες. Αυτό είναι πολύ σημαντική παρατήρηση. Το πακέτο Βασιλεία 3 προβλέπει μια μεγάλη μεταβατική περίοδο. Για να σεβαστούμε αυτές τις απαιτήσει, οι τράπεζες θα πρέπει τα έχουν μέχρι το 2018 και για μερικές κεφαλαίκες επενδύσεις περισσότερο χρόνο. Για να σας δώσω ένα κριτήριο, τα κέρδη των ε, εν λόγω τραπεζών ε, για το 2009 ήταν 96 δις. Η προσαρμογή δηλαδή παίρνει τρία χρόνια κανονικά. Και το 2009 δεν ήταν και από τις καλές χρονιές η Επιτροπή της Βασιλείας προσπάθησε να μετρήσει τον μακροοικονομικό αντίκτυπο των αλλαγών αυτών μέσω μακροοικονομικών προτύπων που βεβαίως και η Τράπεζα της Ιταλίας και η Τράπεζα της Αγγλίας, όλες οι κεντρικές τράπεζες συνέβαλαν να συστάθουν. Το συμπέρασμα ήταν ότι με αυτό το πακέτο ο συνολικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ θα ήταν 0,22% ποσοστιαίες μονάδες στα 25 τρίμηνα μετά που θα ακολουθούσαν τις αλλαγές, δηλαδή 0,03 ε, αναέτος. Αν το συγκρίνουμε με το ΑΕΠ του 2009 θα δείτε πως τα ωφέλη ξεπερνούν το κόστος. Μόνο στην Ιταλία είχαμε 6% απώλειες στο ΑΕΠ τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζουμε ότι το θέμα των μικρομεσαίων είναι πολύ λεπτό γιατί οι μικρομεσαίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη τραπεζική πίστοση και σε ορισμένε χώρες έχουν πιο ευαίσθητη οικονομική κατάσταση, αλλά να θυμίσω σύντομα, το συγγνώμη γιατί φτάσαμε καθυστερημένα σε αυτό το θέμα, τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν ήδη υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση για τις μικρομεσαίες στο πλαίσιο Βασιλεία 2, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Δεύτερον, είναι περισσότερο οι μικρές και μεσαίες τράπεζες που δανείζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτές οι μικρομεσαίες τράπεζες είναι αυτές που θα επηρεαστούν λιγότερο από την μεταρρύθμιση και τρίτον το νέο πλαίσιο δημιουργεί αντικυκλικά εργαλεία μας ζητά να έχουμε ε, φραγμούς για κεφαλαιακούς αλλά και φραγμούς ρευστότητας για να μπορούμε άμεσα να αντιπαρέλθουμε τον περιορισμό της, ε, των δυνατοτήτων όταν μπαίνουμε σε ύφεση. Ούτω ή άλλω όμως αυτά εμείς τα παρακολουθούμε στενά και αν υπάρξει πρόβλημα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων θα επανέλθουμε με αυτά στην Επιτροπή σα. Η Πρόεδρος, ε, συνάδελφοι καθυστερούμε εδώ, τέσσερις επίσημες ερωτήσεις, δεν θα έχουμε χρόνο για έξτρα ερωτήσεις και έχουμε διαργήσει. Παρακαλώ, όχι διπλές ερωτήσεις. Δεν νομίζω πως είναι λάθος του υποψηφίου μας, γιατί έδωσε πλήρες απαντήσεις στις διπλές ερωτήσεις που του θέσατε. Βολφ από το ΕΛΚ, από το Άλντε, συγγνώμη. Μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, οι διάφορες χώρες μέλη αντέδρασαν διαφορετικά στο τραπεζικό τομέα. Άλλοι έκαναν κρατικοποίηση, άλλοι έδωσαν ε, κονδύλια κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ούτως ή άλλως οι διαφορετικές καταστάσεις τρέβλωση του ανταγωνισμού στι χώρε μέλη έτσι και αλλιώ γνώρισαν μια περαιτέρω επιδείνωση και απέχουμε πάρα πολύ από το να φτάσουμε, να επανέλθουμε στην κατάσταση πριν από την κρίση. Ορισμένες ε, ε, χώρες αποφάσισαν να θεσπίσουν κάποιου κάποιους φόρους ε, στις τράπεζες ε, και άλλε μέτρα στρεβλωτικά του ανταγωνισμού. Τι ε, προτίθεστε να κάνετε ούτω ώστε να εξασφαλίσετε να μην υπάρχει αυτή η του ανταγωνισμού και πράγματι να κατατείνουμε προ το στόχο μια πραγματική εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και στον τραπεζικό τομέα. Μια δύσκολη ερώτηση. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι υπήρξαν διαφορετικές αντιδράσεις ε, από τις διάφορες χώρες μέλη. Παρόλο που θα πρέπει να εξάρω το ρόλο της Επιτροπής της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέσπισε κάποια κριτήρια για την ε, κρατική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κρίσης που τουλάχιστον μείωσε το βαθμό διάχυσης ε, αποκλήσεων σε αυτές τις αντιδράσεις των τραπεζών και εξασφαλίσαμε τα πακέτα τα οποία προώθησαν οι χώρες μέλη, αποτέλεσαν και κάποια κίνητρα για την έξοδο από την κρίση και την αποκατάσταση των κριτηρίων ανταγωνισμού εντός της ενίας ευρωπαϊκής αγοράς. Μιλήσατε το αναφερθήκατε στο φόρο επί των ε, τραπεζών ε, ξέρετε ότι η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση με το φόρο αυτό. Η Επιτροπή ε, ε, προέβησε μία ανακοίνωση τον Οκτώβριο και δημοσίευσε ένα έγγραφο εργασίας τον Ιανουάριο εν σχέση με την επίλυση της κρίσης. Και νομίζω ότι εδώ περιλαμβάνονται πολύ σημαντικές και περιεκτικές προτάσεις σε αυτά τα κείμενα. Για παράδειγμα, οι τράπεζες να εισφέρουν σε κάποια ταμεία. Επίσης εξετάζεται η ιδέα ενός ευρωπαϊκού ε, ταμείου. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία επαυλήθηκε από αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι η έκθεση της κυρίας ε, Φερέιρα τόνισε αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, αρκετοί ε, λόγοι να βάζουν στην άκρη τράπεζες εκ των προτέρων κάποια κονδύλια, κάποιους πόρους, που, κάποια κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κρίσης αυτό ε, θα έδινε μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στους επόπτες, ούτω ώστε να αποφύγουμε να ε, κινδυνεύουν τα χρήματα των φορολογούμενων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς, ε, τι μορφή θα προσλάβει αυτό το περιεκτικό πακέτο. Γιατί από τη μία κάνουμε πιο αυστηρές τις απαιτήσει και κεφαλαϊκή επάρκειας, από την άλλη είναι τα κείμενα των G20 που λένε ότι συστηματικά σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να προβλέψουν επιπρόσθετα εργαλεία για να απορροφούν αυτά τα σοκ. Ε, και βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα σύστασης αυτών των ε, ταμείων για την κρίση είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε στο πακέτο αυτό να υπάρχει μια ισορροπία και να υπάρχει μια σωστή αξιολόγηση των επιπτώσεων. Σας ευχαριστώ. Ο Αλφρέντο Μόρα από το ΑΛΚ για τον τρίτο γύρο. Πού είστε, α, κύριε Μάουρο. Σας ευχαριστώ καταρχήν ως Ιταλός ε, για το βαθιά ευρωπαϊκό όραμα και την εικόνα ανεξαρτησίας που δώσατε για την αρχή για την οποία είστε υποψήφιος. Εγώ θέλω να σας υποβάλω το εξή. Η ΕΜΠΑ ενεργοποιείται τώρα που έχει ήδη κραγεί η κρίση και περιμένουμε και ελπίζουμε μάλλον ότι έχει περάσει. Τώρα, αν είχε ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί η ΕΜΠΑ, όταν ξέσπασε η κρίση, τι θα μπορούσε να είχε κάνει και πώς θα είχε συμπεριφερθεί η αρχή. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Μάουρο. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η ΣΕΠΣ... Α, συγγνώμη. Θα τα πω αγγλικά. Εντάξει, δεν θα σας επιτεθώ αν απαντήσετε στα αγγλικά. Η ΣΕΒΣ δουλεύει τώρα σε κάποιους τομείς που αποτελούν την καρδιά της ρυθμιστικής δράσης που έχει ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς αρχίσαμε να δουλεύουμε για τα τραπεζικά κεφάλαια γνωρίζοντας τα προβλήματα για τις διάφορες, διαφορετική μεταχείριση των ε, κεφαλαίων στα διάφορα κατημελία, θυμάμαι καλά ήδη από το 2005. Και ταυτόχρονα αρχίσαμε να δουλεύουμε για το κίνδυνο ρευστότητας. Δυστυχώς, τότε έπρεπε μάλλον μας πήρε κάποιο καιρό να φτάσουμε σε συμπεράσματα, διότι όπως είπα ήμασταν σε πνεύμα συνένεσης, αλλά δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι. Αλλά αυτό που κάναμε, που είναι ήδη στο CRD2, και στις οδηγίες για τη ρευστότητα ήδη καθοδήγησαν προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης. Αλλά έχετε δίκιο ότι υπάρχουν τομείς όπου μάλλον θα είχαμε κάνει περισσότερο αν υπήρχε η ΕΜΠΑ. Δύο τομείς θα είχα να αναφέρω βεβαιότητας. Ήδη το ανέφερα στην απάντηση προς τον κύριο Γκέγκολτ. Η παγίωση των οχημάτων διευθυντικής χρηματοδότησης ήταν καλή η ΕΜΠΑ θα μπορούσε να καταλάβει τις διαφορές εφόσον ε, ε, λειτουργούσε ως σύλλογο, ε, συλλογικό όργανο εποπτικό και να καλύψει τα κενά. Επίσης, αφού είδαμε ότι σε ορισμένες χώρες τα οχήματα ή οι δημοσιονομικοί διαμεσολαβητές κάνουν το ίδιο πράγμα όπως σε άλλες χώρες όπου είναι ρυθμισμένες ε, θα ήταν κάπως ε, χρήσιμο και θα έχει κάπως εμποδίσει ε, τη βλάβη που προκλήθηκε από τον σκεώδη τραπεζικό τομέα. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να ενεργήσουμε στη διάρκεια της επίγουσας ε, ανάγκης. Όταν ξεκίνησε η κρίση, το συζητήσαμε στο ΣΕΠΣΕ και τελικά δεν υπήρξε αρκετή συνένεση για να γίνει πλήρης ερεύνηση, έρευνα μάλιστα, για την έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Και κάτι τέτοιο θα είχε βοηθήσει. Ένα άλλο πιθανό εργαλείο που έχει τώρα η ΕΜΠΑ είναι η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους επόπτες και αυτό θα έχει βοηθήσει τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχουμε ακόμα. Η επόμενη εξ ονόματος των Σοσιαλιστών από την Ελίζα Φερέρα. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντικό που σας ακούσαμε. Και η ερώτησή μου έχει με ένα θέμα το οποίο ήδη αγγίξατε, αλλά θα ήθελα να επανέλθω, που είναι η διαχείριση της πτώχευσης τραπεζών και ιδιαίτερα των ε, συστημικών τραπεζών στην Ευρώπη. Γι' αυτό, γιατί από την αμερικανική άποψη φαίνεται να ε, υπάρχει λύση, ενώ η κατάσταση στην την οποία ζούμε το κόστος δηλαδή για τους ε, φορολογούμενους απαιτεί γρήγορη απάντηση ευρωπαϊκής ε, κλίμακας που να ικανοποιεί και τους πολίτες όπου εμείς ε, ως βουλευτές είμαστε υπόλογοι. Τι ρόλο πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να παίξει η αρχή στην οποία πιθανότητα και ελπίζω θα εκλεγείτε ως πρόεδρος ποια, ποιο ρόλο μπορεί να παίξει όσον αφορά αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση της λύσης για τη διαχείριση των συστημικών κρίσεων. Γιατί αναφέρατε ότι υπάρχουν διάφορα εθνικά προγράμματα που τρέχουν. Άρα λοιπόν έχουμε το, διατρέχουμε το κίνδυνο τη στιγμή που θα ε, βρούμε τη λύση να μην είμαστε σε θέση να την εφαρμόσουμε. Γιατί εδώ μεταξύ εθνικά τα κράτη αυτό που μπορούσαν να έχουν κάνει το έκαναν. Ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι οι αρχές δεν πρέπει ποτέ να βρεθούν σε θέση που δεν θα έχουν επιλογή. Γιατί τότε υπάρχει συστημική, συστημικό λάθος και η μόνη λύση γίνεται η πληρωμή στις τράπεζες. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τρόπους διαχείρισης της εξόδου από τέτοιες κρίσεις. Προηγουμένως, σε προηγούμενη απάντηση, ανάλογης ερώτηση. η Κομισιόν είχε κάνει πολύ λογικές προτάσεις, δηλαδή ότι πρέπει οι αρχές να έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν ορισμένες τραπεζικές δραστηριότητες συγκεκριμένων τραπεζών. Πρέπει να διαθέτουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να ασκήσουν δραστηριότητες που να μην μπορούν να βλάψουν τους καταναλωτές και καταναλώτριες. Ε, ενώ ταυτόχρονα θα πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση των εργαλείων που διαθέτουν οι εθνικές αρχές για να λύσουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, τι ρόλο μπορεί να παίξει η ΕΑΤ συγκεκριμένα. Ένα από τα θέματα που φύγει η Κομισιόν είναι αν οι επόπτες, οι επόπτριες ή άλλες αρχές πρέπει να τα λύνουν αυτά. Εγώ νομίζω οι επόπτες και οι επότεπτριες, γιατί εκείνοι και εκείνες γνωρίζουν καλύτερα ποιες μπορεί να είναι οι σωστότερες τεχνικές λύσεις για επίλυση τέτοιων κρίσεων. Ελπίζω λοιπόν στην νομοθεσία που θα προτείνει η Κομισιόν πριν το καλοκαίρι, ελπίζω, η ΕΑΤ να διαθέτει, να έχει έναν το σωστό ρόλο που πρέπει να παίξει, ιδιαίτερα δε στην αναθεώρηση των ετησίων ε, εργαλείων που θα είναι το κλειδί. Γιατί υπάρχει το άρθρο 18 του κανονισμού για επίγουσες δικαιοδοσίες. Όποτε χρειάζεται να μπορεί η ΕΑΤ να τις συνεργοποιήσει αυτές δεσμευτικά. Σας κατευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Ο Αντιπρόεδρος Μαργκάλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζω με την ερώτηση της κυρίας Φερέιρα. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι η εξής. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα ενιαίο καθεστώς, ευρωπαϊκό καθεστώς για, τα, για τις διασυνοριακές ευρωπαϊκές τράπεζες ε, θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις για αυτού του είδους τις οντότητες. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαία μια ειδική ευρωπαϊκή εποπτεία για αυτές τις οντότητες, για αυτούς τους οργανισμούς. Πιστεύετε ότι, υπάρχει, ότι είναι αναγκαίος ένας μηχανισμός επίλυσης της κρίσης για, αυτές τις, για αυτούς τους οργανισμούς και πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό ταμείο σταθεροποίησης, διαφορετικό από τα εθνικά ταμεία για αυτές τις διασυνοριακές ε, τραπεζικές οντότητες ή διασυνοριακά τραπέζια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαρθία Μαργκάλιο και θα ήθελα επίσης να σε ευχαριστήσω για την εργασία που κάνατε στα επίπεδο της ε, ρύθμισης που πραγματικά ενισχύει το ρόλο της ε, ΕΜΠΑ, της ΕΑΤ. Ξέρω ότι στην έκθεση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζεται το ενδεχόμενο της ενίσχυσης του ρόλου της ΕΑΤ στην άμεση εποπτεία των διασυνοριακών ομίλων. Επίσης, ε, ε, όσον αφορά ε, ένα, μια ενότητα επίλυσης της κρίσης σε περίπτωση, σε περίπτωση κρίσης αυτών των διασυνοριακών ιδρυμάτων. Εγώ θα εργαστώ βεβαίως ε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου και πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη παρόλα αυτά για ενιαία εργαλεία επιπρόσθετα προς τα εθνικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των κρίσεων των εθνικών ρυθμιστών. Ήδη στη ρύθμιση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να λειτουργήσει σαν διαμεσολαβητής εάν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των εθνικών αρχών. Και εγώ θα περίμενα εάν υπάρχει μια συνάντηση ε, μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, εγώ θα ανέμενα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να λάβει μέρος σε αυτή την ε, συνάντηση ούτε ώστε να εισφέρει για τη διευθέτηση των διαφορών ως ανεξάρτητη αρχή. Εάν υπάρχει ενδεχομένω μια κίνηση προς, μια, προς ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επίλυσης των Κρίσεων, ιδέα την οποία εγώ θεωρητικά υποστηρίζω τότε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών θα είναι καθοριστικός ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση, δηλαδή τα χρήματα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό το ταμείο να αξιοποιούνται προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τις εξαιρετικά περιεκτικές τις απαντήσεις. Ε, δεν έχουμε χρόνο για επιπλέον ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν η ακρόαση και θα έχουμε τώρα μια συζήτηση και κλεισμένων των θυρών αποκλειστικά μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας και όσοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν σε αυτή τη συνεδρίαση παρακαλούνται να εγκαταλείψουν την αίθουσα. I, I think this is an opportunity for some quick...